Welcome to the meeting. <clears throat> All the languages are available. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Όλες οι γλώσσες εκτός από κροατικά και μαλτέζικα υπάρχουν στη διερμηνία. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι έχουμε δύο ομάδες επισκεπτών. Ο κύριος Χαβιέρ Λόπες καταρχήν έχει μια ομάδα 30 σοσιαλιστές από την Καταλωνία και θα παρακολουθήσουν από τις 11.30 την ε, συνεδρίασή μας. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ επίσης 21 άτομα έχει μαζί της μια ομάδα επισκεπτών που θα παρακολουθήσουν το θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική από τις 11 και 4 ως τις 12.30. Κατόπιν έχουμε και μια άλλη ομάδα επισκεφτών που έχει καλέσει ο κύριος Φουντούλης. Πρόκειται για φοιτητέ ε, πολιτικών επιστημών οι οποίοι θα παρακολουθήσουν από την αρχή, δηλαδή από τώρα, την συνεδρίασή μας. Όλοι όσοι είστε εδώ λοιπόν σας καλωσορίζουμε. Και βεβαίως και όλοι όσοι δεν έχουν έρθει ακόμα τους καλωσορίζουμε επίσης. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω όσον αφορά τη συνεδρίες μας της 17ης Νοεμβρίου. Είχαμε προσκληθεί και εγώ μάλιστα σαν προεδρεύουσα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ήμουν προσκεκλημένη, καθώς και η κυρία Κούνεβα, ο κύριος Μέσεριτς, η Μαρία Ροτρίγκες και ο Βάντεν Κέντελερε και άλλοι ήταν προσκεκλημένοι, ήμασταν όλοι παρόντες, ίσως ξέχασα μάλιστα και κάποιους από τους ε, παρόντες της συνεδρίας κανείς. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη κατά την άποψή μας, καθότι τα θέματα που συζητήθηκαν είναι θέματα ε, πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για μας. Και μάλιστα πήραμε το λόγο και συμμετείχαμε σε πολλές από τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα. Θα ήθελα να περάσω τώρα στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται για τον ε, τριμερή διάλογο. Θα ήθελα καταρχήν να δω ποιος είναι εδώ έτσι ώστε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Άγνες, θέλω να σου δώσω το λόγο. Κάτσε γρήγορα. Οι συνεδριάσεις που έγιναν καταρχήν η πρώτη ήταν στο Στρασβούργο στις 13 Δεκεμβρίου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική συνεδρίαση όσον αφορά τα αποτελέσματα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση εκκίνησης. Η επόμενη θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες και στις 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες επίσης, αλλά και στις 13 ε, Δεκεμβρίου εκ νέου στο Στρασβούργο. Δεν ξέρω βέβαια, αν ε, μπορούμε να είμαστε απολύτως αισιόδοξοι. Ο, η πρώτη συνάντηση τριμερούς διαλόγου ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι στις 13 Δεκεμβρίου μπορούμε να ελπίζουμε σε θετικά αποτελέσματα. Να δώσω το λόγο στην γυρία Γιονγκέριος, έτσι ώστε να μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής ε, της πρώτης συνάντησης τριμερούς διαλόγου, καθώς και των ε, προτάσεων των σκιωδών εισηγητών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήδη δώσατε κάποιες από τις ε, πληροφορίες που ήταν ε, σημαντικές. Και εγώ θεωρώ ότι ξεκινούμε από ένα θετικό, θα έλεγα, αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο βεβαίως να βρεθεί κοινό έδαφος, υπάρχουν πολλές ε, διαφορετικές προτάσεις, αντιπροτάσεις και βεβαίως και εμείς έχουμε και τη δική μας ε, εντολή για τη συζήτηση αυτή. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η πρώτη συνάντηση τριμερούς διαλόγου για να εξηγήσουμε ποια είναι τα θέματα που εμείς θεωρούμε ουσιαστικά. Το Συμβούλιο επίσης και η Επιτροπή έχει τις δικές της θέσεις, τα δικά της κεντρικά σημεία. Είναι πλέον σαφές σε όλους ποιες είναι οι θέσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ και ο συνεισηγητής έρχεται, θα μπει στην αίθουσα από στιγμή σε στιγμή. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που μας ε, υπέβαλε το Συμβούλιο Έχουμε εντοπίσει τα θέματα αυτά, τα οποία θα αποτελέσουν το επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη διάρκεια αυτών των τριών συναντήσεων, όπως αναφέρατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, αυτές τις τρεις ημερομηνίε που έχουν προβλεφθεί. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα της Προεδρίας του Συμβουλίου και φυσικά και οι αντιπρόσωποι της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει έχουν το θέμα αυτό πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους. Αν λοιπόν αποτύχει η Εστονική Προεδρία να ολοκληρώσει την ε, συζήτηση αυτή, πιστεύω ότι η επόμενη Προεδρία θα το ολοκληρώσει. Τουλάχιστον είναι πολύ ε, σημαντικό το θέμα για αυτούς όπως έχουν ανακοινώσει. Είμαι, αν θέλετε, αρκετά θετικά διατεθειμένη και πιστεύω ότι υπάρχουν ελπίδες να βρεθεί λύση. Υπάρχουν σχόλια. Καλωσορίζω όσους μπήκαν στην αίθουσα. Καλωσορίσατε. Η επόμενη συνάντηση των σκιωδών για το θέμα αυτό είναι στις 27 Νοεμβρίου στις 8 το πρωί. 8 με 9. Όχι, λέει Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη. Είναι από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Αργά το απόγευμα δηλαδή. Εντάξει. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ξέρετε ότι όσον αφορά την Επιτροπή Μεταφορών έχουμε μία διαμάχη, μία διαφορά όσον αφορά το θέμα των ε, χερσαίων μεταφορών, των οδικών μεταφορών και Γνωρίζετε φαντάζομαι το θέμα. Αυτό μπορείτε να μας ενημερώσετε. Πρόκειται για το άρθρο 54 και εδώ θα πρέπει να αποφασίσουν τα αρμόδια μέλη της Επιτροπής. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έγκριση των πρακτικών της 16ης Οκτωβρίου και της 19ης Οκτωβρίου του 2017. Εγκρίνονται τα πρακτικά και θα περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για το θέμα που αφορά το Europass. Εδώ ε, στις 9 Νοεμβρίου Έλαβε χώρα η δεύτερη συνάντηση τριμερούς ε, διαλόγου. Ο κύριος Μάνα θα μας κάνει μια σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων και θα μας παρουσιάσει και τα επόμενα σημεία. Κύριε Μάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι το Europass μπορεί να γίνει μια μάρκα εναερίων μεταφορών στην Ευρώπη προκειμένου περί δεξιοτήτων και προσόντων, αν φερθούμε σωστά. Είναι εθελοντικός μηχανισμός και ήδη έχουμε συμφωνήσει σε πολλά. Στις 9 Νοεμβρίου, στο κτίριο του Συμβουλίου εδώ στις Βρυξέλλες, μπορέσαμε να μιλήσουμε για το τι δέον γενέσθε Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Καταρχήν ευχαριστήσω θερμά τη γραμματεία. Η προετοιμασία τους ήταν πολύ καλή. Αλλά και οι τεχνικές ομάδες, τόσο της Κομισιόν όσο και του Συμβουλίου, ε, προχώρησαν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ομαδικό πνεύμα που δεν το βλέπουμε τόσο συχνά σε χώρες όπως τη δική μου για παράδειγμα τώρα τελευταία. Υπάρχουν διάφορες ανάγκες για συγκεκριμένους ορισμούς. Εκεί προχωρήσαμε καλά. Μπορώ να πω στα μέλη της Επιτροπής ότι έχουμε ένα κοινό, η Επιτροπή ε, Πολιτισμού και Απασχόλησης συνεργάστηκαν. Συμφωνήσαμε σε 72 σημεία που είναι ήδη πολλά είναι τα δύο τρίτα δηλαδή. Καταφέραμε πολλά. Προβλήματα υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τις δεξιότητες. Εδώ υπάρχουν πολλές διαφορές και μεταξύ των ομάδων. Οπότε στην τέταρτη συνάντηση των Σκιωδών στις 14 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο ε, διαπιστώσαμε ότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει. Οπότε παίρνει παράταση το θέμα. Και εδώ όμως υπάρχει βούληση για συμβιβασμό. Αν ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο εμπόδιο, τότε θα έχουμε προχωρήσει πολύ σημαντικά. Το κλίμα ήταν καλό, μπορούμε να το ακούσουμε και από την πρόεδρο που ήταν εκεί, οπότε υπάρχει πρόθεση προσέγγισης, υπάρχει βούληση για καλό αποτέλεσμα. Μετά έχουμε τον τριμερή διάλογο στις 7 Δεκεμβρίου ο επόμενος. Δεν ξέρω αν θα είναι ο τελευταίος, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα έχουμε προχωρήσει. Και προηγουμένως έχουμε και μια συνάντηση των σκιωδών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και αν καταλήξουμε και συμφωνήσουμε με Συμβούλιο και Κομισιόν, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, αυτή την ε, ε, νέα ευρωπαϊκή μάρκα εναερίων μεταφορών. Πάμε καλά, υπάρχει συμβιβαστικό πνεύμα και ευχαριστώ που μπόρεσα να δώσω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Μαν. Άλλος κανείς θέλει να μιλήσει για το Europass. Ξέρουμε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Όλοι, ακόμα αυτοί που δεν το γνωρίζουν από κοντά το θέμα. Ε, γίνεται συζήτηση όπως είπατε κυρία Μάν και με τους κοιόδης και ε, ένα σημαντικό θέμα είναι οι ε, δεξιότητες και η σχετική πληροφόρηση γιατί πολλές φορές δίνονται πληροφορίες σχετικά με επαγγέλματα και δεξιότητες που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Εμείς κάνουμε προσπάθειες προς μια απόφαση που θα βρει όλους σύμφωνους σχετικά με το πώς θα συνεχίσουμε και ελπίζω ότι όταν γίνει στις 7 Δεκεμβρίου ο τριμερής διάλογος θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και να είναι όντως ο τελευταίος τριμερής. Δεν βλέπω να ζητεί άλλο το λόγο. Οι δεξιότητες όπως γνωρίζουμε ε, αποκτούν ε, πολύ μεγάλη σημασία τα επόμενα χρόνια. Ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει κανείς από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, η κυρία Κραμπ. Παρακαλώ, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Λέγομαι Κράμπ, είμαι από την ε, μονάδα δεξιοτήτων και προσόντων και εξειδίκευσης. Όπως είπε και ο κύριος Μαν, πιστεύω ότι υπάρχει θετική πρόοδος, ένα κλίμα επικοδομητικό. Από την Κομισιόν εμείς ε, συμμετέχουμε πάρα πολύ στις προπαρασκευαστικές εργασίες σε επίπεδο τεχνικών ομάδων και οι εμπλεκόμενοι μας πιέζουν, δηλαδή και από την αγορά εργασίας, οι εμπλεκόμενοι και από την εκπαίδευση και από την κατάρτιση, προσβλέπουν σε εμά να μπορέσουμε να ε, εξυγχρονίσουμε το Europass και όπως είπε και ο κύριος Μαν, οι συζητήσεις φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο. Και προχωρούμε γρήγορα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Η πρόταση συζητείται εδώ και αρκετό καιρό στο Συμβούλιο πρέπει να πω και γνωρίζομαι ότι οι εμπλεκόμενοι ανυπομονούν να δουν βελτίωση στις υπηρεσίες αυτές που θα, εξυπηρετήσουν και την αγορά εργασίας αλλά και την εκπαίδευση και τις σπουδές. Είμαστε λοιπόν σε καλό δρόμο προς μια συμφωνία και νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, άντε τους επόμενους μήνες, θα συμφωνήσουμε. Ο κύριος Μαν θα έχει τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πράγματι κινηθήκαμε ο ένας προς την κατεύθυνση του άλλου, είναι καλό αυτό, έχουμε συμβιβαστικό πνεύμα και αν ελπίζω να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό και θα συνδέεται με αύξηση της κινητικότητας σε τελευταία ανάλυση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να Δύο λεπτά σας δίνω να βρείτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες και μετά πάμε στην ψηφοφορία.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 Λοιπόν, όλοι έχετε εισαγάγει τις κάρτες στο μηχάνημα, αρχίζουμε. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμοποίηση. Το πρώτο είναι τομέας Λιανικής ε, στη Φιλανδία. Άρχεται η ψηφοφορία. And Πέρας. Δεκτό με 30 ψήφους υπέρ. Το άλλο θέμα κινητοποίησης του Ταμείου είναι η... ο τομέας Λιανικής στην Ελλάδα, στην Αττική. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας πάλι δεκτό με ψήφους υπέρ 30. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Καθυστέρησα να ψηφίσω. Ήθελα να ψηφίσω υπέρ και εγώ. Σημειώστε το. Εντάξει. Δεν κάνει διαφορά βέβαια ουσιαστική, το ξέρω αυτό. Πάντα έχει διαφορά. Πάντα η ψήφος κάνει διαφορά. Ε, η διατάξη εσές υπέρ, κατά... Α, όχι πρέπει να είναι και αυτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τις διατάξεις ESF. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28 ψήφοι υπέρ, γίνεται δεκτό. Ε, οπότε έχουμε τα αποτελέσματα των τριών ψηφοφοριών. Μα είμαστε στο μέσο της ψηφοφορίας. Ναι, κυρία Φουντούλη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μικρόφωνο, κύριε Φουντούλη. Δεν δουλεύουν κάποια μηχανήματα, κύριε Πρόεδρε. Can someone help, Mr. Ε, μπορεί κάποιος να βοηθήσει τον κύριο Φουντούλη, ίσως να αλλάξετε ε, έδρανο. Τώρα είναι εντάξει. Ε, πρέπει να ξαναψηφίσουμε για το Omnibus, για τις διατάξεις ESF. Λοιπόν, επαναλαμβάνομαι την ψηφοφορία. Κανονισμός, ε, Omnibus, διατάξεις ESF, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 32 ψήφοι υπέρ. ε, μπορείτε να πάτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο μηχάνημα. Προχωρούμε στην επόμενη. Γιάση GF Feed, οι σχετικές διατάξεις. Ποιοι είναι υπέρ, ονομαστική είναι η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Και ε, ο κανονισμός με τις τέσσερις ε, στήλες, ο κανονισμός όμνιμπους το σχέδιο, πέρας. Υπάρχει αποτέλεσμα. Υπάρχει 32 ψήφοι υπέρ. 2 κατά, 6 αποχές. Προχωρούμε.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 Ε, αρχίσαμε ήδη την ψηφοφορία. Όσοι ήρθαν καθυστερημένα έχουν ελάχιστο χρόνο να καθίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Αρχίζουμε. Ε, έκθεση Φάλτος Φερμέγιος. Περιμένουμε το κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, έκθεση Λόπες Μπερμέγιο. Υπέρ της έκθεσης Εσείς είστε κατά. Ε, ε, αν ψηφίσετε υπέρ, απορρίπτετε την έκθεση. Αν γίνει δεκτή, όλες οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν. Υπέρ. Κατά. συγγνώμη, τι ψηφίζουμε, έχουμε μπερδευτεί, δεν έχουμε καταλάβει. Ποια έκθεση ψηφίζουμε. Την, ε, το τεστ αναλογικότητας. η νομοθετική ε, ε κατοχήρωση των επαγγελμάτων. Ψη, δοκιμή αναλογικότητας πριν από την έκδοση νέων ε, ε, αποφάσεων. Έκθεση ε, Λόπες Μπερμέγιο. Έλεγχος αναλογικότητας. Αυτό το ψηφίσαμε. Συνεχίζουμε να ψηφίζουμε. Θα απορρίψουμε το σύνολο και πάμε στην τροπολογία 1. Αποσύρθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ ελέγχουμε την συμβιβαστική αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 31 ψήφι κατά. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, καταπίπτει 89. 95. Ποιος είναι υπέρ. 95. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ελέγχουμε την 99, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται 25 υπέρ. 101 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε τη συμβιβαστική 2, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, η συμβιβαστική 2 εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 111, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίφθηκε με 23. 112. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά ελέγχουμε την 112. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Με 31 ψήφους κατά. 113 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική β, συγγνώμη, 3, συμβιβαστική 3, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε τη συμβιβαστική 3, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται με 33 ψήφους κατά. Συμβιβαστική Β, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την Β, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. εγκρίνεται με 34. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 107. Ψηφίζουμε την 107. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την συμβιβαστική 5. Αρχή της ψηφοφορίας. Συμβιβαστική 5. Τέλος. Εγκρίνεται με 25 υπέρ. Συμβιβαστική. Λάθος. Τροπολογία 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 139 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε την 139 αρχή της ψηφοφορίας τέλος απορρίπτεται με 34 κατά 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, ελέγχουμε την 7, συμβιβαστική 7. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική, όχι. Λάθος. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 159 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Η τροπολογία 159 ψηφίζουμε την 160. Κατά, αποχές, ελέγχουμε την 160, αρχή της ψηφοφορίας, τέλος, εγκρίνεται με 22 υπέρ. Τροπολογία 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 162 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την συμβιβαστική ε, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται με 36 πέρα. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω εγκρίνεται, ελέγχουμε την 8, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, εγκρίνεται με 25 υπέρ. Περνάμε στην συμβιβαστική εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τροπολογία 187 και 188 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε όμως την 190 190 αρχή της ψηφοφορίας Τέλος. 23 υπέρ 23 κατά. 196 και 198 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. 196 και 198 Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται με 33 ψήφους κατά. 200. Τροπολογία 200. Και 301 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, εν... απορρίπτεται. Με 32 ψήφους κατά, λέει η πρόεδρος. 202 και 204 είναι ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 203 έχει αποσυρθεί. 206 και 207 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 206 και 207 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτονται με 32 ψήφους κατά. Μπορείτε να σηκώνετε τα χέρια σας λίγο πιο διακριτά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή την αίθουσα να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις ψήφους. 233 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 209 και 210 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 11 αποσύρθηκε. 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 214. 15 και 16 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.15. Να ελέγξουμε για τις 2.14 και 2.16. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. 215 τροπολογία απορρίπτεται. Συγγνώμη, καταπίπτει. Και πάμε τώρα, λέει πρόεδρο στην τροπολογία 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ...224 υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνεται... ...225 υπέρ... ...όχι τώρα δεν καταπίπτει... ...υπέρ ξαναλέει η πρόεδρος υπέρ... ...κατά αποχές απορρίπτεται θα έλεγα η 225 συμβιβαστική πρόταση 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική 10 παρακαλώ πέρα στις ψηφοφορίας εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 11. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας για τη συμβαστική 11. Απορρίπτεται με 32 ψήφους κατά. Μετά έχουμε και τις επόμενες, λέει πρόεδρος. 234, 35 και 37. Ομού, μαζί. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Εγκρίνονται. Συνεχίζουμε. Πάμε στη συμβαστική πρόταση F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το F. Ωραία. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Πάμε στην επόμενη σελίδα, σελίδα 13, συμβαστική 13, υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 13. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 13. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Με 33 ψήφους κατά. Συμβαστική 14. Όχι, ένα το λέει πρόεδρο. Θα πρέπει να ψηφίσουμε μία προς μία τις επόμενες τροπολογίες. Πάμε λοιπόν στην 248. 248 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για 249. Ωραία. Καταπίπτει όμως, γιατί υπερψηφίσαμε τη 248, λέει η Πρόεδρος. Yeah. It has fallen, amendment 249. Η 249 καταπίπτει. We, we rejected Απορρίψαμε τη 248 λέει ο πρόεδρος το οποίο σημαίνει ότι αυτή εδώ η 249 καταπίπτει. Οπότε πάμε στη 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 14. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με 36 ψήφους κατά. Πάμε στην 253 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την συμβαστική 15. Άρχεται. Πέρας. απορρίπτεται με 35 ψήφους κατά. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές νομίζω θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 16 άρχεται πέρας απορρίπτεται με 31 ψήφους κατά Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει πρόεδρος. Όχι. Ε, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τότε για τη συμβαστική 17. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 36 ψήφου. κατά λέει πρόεδρο, συγγνώμη. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. αποχέ. εγκρίνεται. It's impossible to see in this room when you're spread out. Δεν μπορώ να σα βλέπω όλου. Είστε σκορπισμένοι στην αίθουσα. 18. Για 18 συμβαστική. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λέει η πρόεδρος. We τη ψηφοφορία. Το ίδιο αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρο. Απορρίπτεται με 36 ψήφου. κατά. Πάμε στη 19. Συμβαστική 19. Να μα ψηφίσουμε ωραία. 19. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Thank you. Ευχαριστώ. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μια ερώτηση, Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπήρχαν εδώ σε αυτές τις συμβαστικές και κάποιες υποτροπολογίες. Αν απορριφθεί μια συμβιβαστική, πρέπει να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες οι οποίες στην 18 παραδείγματος χάνει τη συμβαστική. Δεν το κάνετε αυτό. The reason why we don't do that. Ο λόγος για τον οποίο δεν το κάνουμε είναι επειδή είναι ταυτόσιμες οι τροπολογίες αυτές είναι ταυτόσιμες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν ψηφίζονται. Δεν τίθεται σε ψηφορία δηλαδή, λέει πρόεδρος. Να ψηφίσουμε όμως για την 276. 276. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμβιβαστική η 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, δεν θέλετε, ωραία, θα ψηφίσουμε τότε ηλεκτρονικά για την συμβαστική 22. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 22 απορρίπτεται με 37 ψήφου κατά. Τροπολογία 280 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 280 θέλετε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για 280. Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά. 281. Δεν ψηφίζουμε 282. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για 282. So the vote And the vote is now closed. Πέρας τώρα. Απορρίπτεται. 283. Υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για 283. πέρα τη ηλεκτρονική για τη 283. Ναι, ακριβώ το ίδιο αποτέλεσμα όπως πριν, λέει η πρόεδρος. 284 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ it will don't θα πάμε στη 282 λέει ο Πρόεδρος. 242, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε για τη συμβαστική, αλλά η 242. 242 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Να αλλάξουμε. Ωραία, 242 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 243. Την ψηφίζουμε 243, ρωτάει πρόεδρος. Ωραία, 243. Υπέρ, υπέρ 243. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 244 δεν ψηφίζουμε. Πάμε στο 287. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για την 287 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες για την 287 απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 200 για συγγνώμη για την 23 συμβαστική 23 συμβαστική 23 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία Πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη συμβαστική 23 απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά λέει πρόεδρος συμβαστική age υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική Age. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. Επόμενη τροπολογία. 296. 296 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 298 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 298. Άρχεται για την 298. Η ηλεκτρονική ψήφος. Πέρας για την 298 απορρίπτεται. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. Πάμε στη 297. 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 302 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 302 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 28 Ψήφου κατά 301 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 303 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται τροπολογία 304 υπέρ κατά Αποχέ. θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 304 άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται, λέει πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 306. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, το ίδιο αποτέλεσμα όπω έλεγα, λέει πρόεδρος. 307. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 308. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στα εκτιμώντας τροπολογία 3 στα εκτιμώντας 1 τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 8 άρχεται Πέρας τώρα της ηλεκτρονικής πληροφορίας απορρίπτεται με 26 ψήφους κατά. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική. Όχι. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 9. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 9. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Να ξαναψηφίσουμε λέει Πρόεδρο για την 24. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ της 24. Κατά. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 28 ψήφους υπέρ. Τροπολογία. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Καταπίπτει. 20. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο 8. Τροπολογία σκέψη 8. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Άι υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την Άι Άρχεται. Πέρας. Και εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Συμβαστική J. Όχι, λέει πρόεδρος. Πάμε στην τροπολογία 27. 27, τροπολογία 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τα 32. Άρχεται η ψηφορία. Τέλος. Απορρίφτεται. Με 36 κατά. Και τώρα περνάμε στην 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35. Να ψηφίσουμε και τη 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και με την κάπα, συμβιβαστική κάπα, τι κάνουμε, λέει η πρόεδρος. Ψηφίζουμε την κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία για την συμβιβαστική 28. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 28. Συμβιβαστική έλα, λάμδα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 50 αρχή της ψηφοφορίας τέλος Απορρίπτεται η 50. 27 κατά. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 56. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 57, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 58, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ελέγξουμε την 29 Υπέρ. Συγγνώμη, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος της ψηφοφορίας. Είστε έτοιμοι? Όχι, ε, λέει η πρόεδρος. Κάποιος επιπλέον έχει ψηφίσει από το ΕΛΚ. Τώρα όμως είναι εντάξει. Απορρίπτεται. 27 ψήφοι κατά. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 68 αρχή της ψηφοφορίας τέλος εγκρίνεται 69 καταπίπτει. 71 Υπέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 74. Τέλος. Απορρίπτεται. 72 κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 30. Αρχή της ψηφοφορίας, τέλος, απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Συμβιβαστική νη, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την συμβιβαστική νη. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική για την 87, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 87 ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. Με 26 ψήφους υπέρ. 88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του τροποποιημένου κειμένου. Αρχή της ψηφοφορίας. Αρχή της ψηφοφορίας για το σύνολο του κειμένου. Τέλος. Απορρίφθηκε. τελικά απερίφθη, αλλά παρόλα αυτά ευχαριστούμε τον εισηγητή για την ε, δουλειά του. Is this uh, where now? This is Uh, λοιπόν, αγαπητοί μου, προχωρούμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ηλεκτρονική κάρτα. Όσοι δεν θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση αυτή μπορείτε να αποχωρήσετε. Και εμείς οι άλλοι θα μιλήσουμε για την ηλεκτρονική κάρτα. Λοιπόν, μισό λεπτό θα περιμένουμε και μετά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Όσοι πάρετε τη λάθος απόφαση να φύγετε και να μην ακούσετε τη συζήτηση για την ηλεκτρονική κάρτα, φύγετε τώρα. Είμαστε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή ε, ηλεκτρονικής κάρτας ευρωπαϊκών υπηρεσιών και οι συναφείς διοικητικές ευκολίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ε, τροπολογίες, τους 104 συνολικά. Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην πρόταση αυτή νομίζω. Από τους συναδέλφους, τους σοσιαλιστές και τους πρασίνους έχουμε πρόταση απόρριψης της πρότασης της Κομισιόν για την κάρτα. Γίνεται και σε άλλες επιτροπές αυτό, γιατί είμαι σκιώδης και αλλού. Άλλοι συνάδελφοι όπως εγώ πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιες σοβαρές ανησυχίες βέβαια εν ώψη αυτών των προτάσεων, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιωθούν από μας αυτές οι προτάσεις για να υποστηριχθούν στο τέλος. Εις ό,τι αφορά την απόρριψη της πρότασης, ο βασικός λόγος είναι ότι ο σκοπός ήταν να βελτιωθούν οι διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών, αλλά κάποιοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι δεν πρόκειται για την ελεύθερη διακίνηση, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά η έλλειψη των μέτρων ελέγχου ε, επί των εταιριών που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη εποπτεία, επιτήρηση, μέτρα ελέγχου, ούτω ώστε οι εταιρείε να συμμορφούνται προς τους κανόνες του κράτους μέλους υποδοχής. Και αν μπορώ να συνοψίσω την άποψη αυτή σε μια πρόταση θα ήταν ότι από τώρα το σύστημα δεν λειτουργεί καλά, όχι τώρα το σύστημα δεν λειτουργεί καλά και αυτό σημαίνει ότι ε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Άλλοι συνάδελφοι και εγώ μαζί τους πιστεύουμε ότι ενώ η πρόταση αυτή έχει σοβαρούς περιορισμούς παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι Αξίζει να συζητήσουμε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για να δούμε αν υπάρχει κοινό έδαφος και αν στο τέλος θεωρήσουμε ότι η πρόταση αυτή όντως θα βελτιώσει την κατάσταση σχετικά με κάποια από τα θέματα που έχουν τεθεί. Το πρώτο που θέλω να πω, θα τα πω σύντομα, γιατί ε, ενδιαφέρει να δούμε τις διαφορετικές αποχρώσεις και το σκεπτικό το διαφορετικό. Δύο λόγια από μένα. Για το θέμα του κατασκευαστικού τομέα, όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι προτείνουν την εξαίρεση του τομέα αυτού από την πρόταση. Αυτή είναι η γενική άποψη που επικρατεί. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αποχρώσεις και εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρχει δυσκολία να βρεθεί συμφωνία. Το θέμα της ασφάλισης είναι λίγο πιο σύνθετο. Κάποιοι θέλουν να εξαιρεθεί τελείως, άλλοι συνάδελφοι θέλουν ε, να φύγει το υποχρεωτικό σκέλος της ασφάλισης, αλλά να υπάρχει υποχρεωτική ενημέρωση για την ασφάλιση. Αλλά κοιτάζοντας τις τροπολογίες και πάλι, ελπίζω ότι υπάρχει ε, δυνατότητα να βρούμε κοινό έδαφος για το θέμα των διατάξεων για την ασφάλιση. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που θέλουν να δώσουν μεγαλύτερο λόγο στο κράτος μέλος υποδοχής και ειδικότερα να διασφαλίσουν ότι όλοι οι, όλες οι πληροφορίες θα επαληθεύονται σωστά και θα εξακριβώνονται. Αυτή είναι καλή προσέγγιση γιατί αυτό σημαίνει είναι ότι δεν πάμε να διορθώσουμε εκ των υστέρων σφάλματα, αλλά από την αρχή θα έχουμε ένα σύστημα σωστό και θα αρχίζουμε με στιβαρές διατάξεις, για τις οποίες θεωρούμε ότι ε, θα εξασφαλίσουν ακριβείς πληροφορίες. Τώρα, για την μονοθυριδική υπηρεσία και εδώ υπάρχουν πολλές τροπολογίες και μπορεί να γίνει πολλή συζήτηση, πολλές προτάσεις για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής κάρτας και τη μεγαλύτερη ευελιξία εις ό,τι αφορά τις προθεσμίες. Εγώ πιστεύω ότι οι προθεσμίες που προτείνονται από την Κομισιόν είναι πάρα πολύ σφιχτές και οι περισσότεροι συνάδελφοι πιστεύουν το ίδιο σχετι... Ε, προκειμένου περί της ε, παράτασης της προθεσμίας. Ένα θέμα επίσης άλλο ε, είναι οι εγκρίσεις. Υπάρχουν και κάποιες άλλες θετικές προτάσεις που μπορώ να στηρίξω και ορισμένες προτάσεις σχετικά με τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν σχετικά με την εκτελεστική πράξη. Σε σχέση ε, ε, με την αρχική πρόταση της Κομισιόν δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμε τις εκτελεστικές πράξεις που προτείνονται εκεί γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και ασάφεια. Αυτά. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να βελτιώσουμε το, την πρόταση. Αυτό είναι το δικό μου πνεύμα. Με αυτό το πνεύμα αρχίζω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Ο κύριος Κοχ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Θα είμαι σύντομος. 104 είναι συνολικά οι τροπολογίες για την πρόταση της ηλεκτρονικής κάρτας παροχής υπηρεσιών. Από αυτές τις 104, 43, οι μισές δηλαδή περίπου, κατατέθηκαν από το ΕΛΚ. Αυτό δείχνει ότι ως ομάδα εμείς το ΕΛΚ βλέπουμε με κριτικό μάτι το κείμενο. Παρ' όλα αυτά όμως αποφασίσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτή την ηλεκτρονική κάρτα και να εργαστούμε για να βελτιωθεί το κείμενο. Ε, δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσει η ψηφιοποίηση και δεύτερον, να μειωθεί η γραφειοκρατία. Η ηλεκτρονική αυτή κάρτα ανοίγει ένα τέτοιο παραθυράκι. Ε, γι' αυτό ε, χαίρομαι για τις συμβιβαστικές που θα καταρτιστούν και για τη συνάντηση των σκιωδών την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γιονγκέριος. Ευχαριστώ. Χρησιμοποιώ το κείμενο της κυρίας Ρέγνερ που είναι σκιώδης και δεν μπόρεσε να έρθει και έχει καταγράψει πέντε σημεία ε, για τα οποία πρέπει να απορριφθεί η πρόταση. Πρώτον, οι προτάσεις ε, εισάγουν από την πίσω πόρτα την αρχή της ε, χώρας καταγωγής και οι αρμοδιότητες του κράτους υποδοχής μεταφέρονται στο κράτος ε, καταγωγής. Ε, έτσι υπονομεύονται οι αρμοδιότητες ε, της χώρας υποδοχής και ο κοινός παρανομαστής πέφτει αισθητά. Προσαρμοζόμαστε στις χειρότερες συνθήκες. Επίσης, η κάρτα αυτή θα διευκολύνει ε, λέμε ε, εταιρείε να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά. Η ε, ψεύδο αυτοαπασχόληση όμως δεν θα μειωθεί, αντίθετα μπορεί να αυξηθεί, να παρουσιάζονται δηλαδή ως αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι που μπορεί να δουλεύουν για μια, να είναι αποσπασμένοι σε μια εταιρεία. Επίσης το forum shopping θα προαχθεί, δηλαδή επιλογή του ευνοϊκότερου δικαστηρίου και αυτό δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για dumping, μισθολογικό, απάτες και αδήλωτη εργασία. Η πρόταση τρίτων δεν παρουσιάζει ε, αξιόλογα μέτρα ελέγχου ε, στη χώρα υποδοχής και αυτό μπορεί να υπονομεύσει ε, γενικότερα τους ελέγχους και το έργο των επιθεωρητών εργασίας. Τέταρτον, η κάρτα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποσπασμένους. Έτσι δημιουργείται μεγάλη κοινωνική αβεβαιότητα. Ενώ κλείνουν τα παραθυράκια για τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους, θα ανοίξουν μέσα από την κάρτα νέα παραθυράκια τα, και αυτό αντιφάσκει προς τη θέση του Κοινοβουλίου για την απόσπαση εργαζομένων. Πέμπτον και τελευταίον, η ε, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου δεν δίνει καμία προστιθέμενη αξία. Αντίθετα, οι εταιρείε και οι απασχολούμενοι τους θα πάθουν σημαντική ζημιά λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού που θα προκύψει. Γι' αυτό η σκιώδης εισηγήτρια ζητεί να απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν και θα προσθέσω και εγώ κάτι προσωπικό δικό μου. Σε δημόσιες συναντήσεις η ίδια η Κομισιόν λέει και παραδέχεται ότι υπάρχουν μεγάλες αδυναμίες στην πρόταση αυτή. Ας τη βοηθήσουμε στέλνοντας την πρόταση πίσω στην Κομισιόν να αξιοποιήσουμε το χρόνο για να σκεφτούμε ξανά και εμείς και εκείνοι πάνω στην πρόταση αυτή και να υποβάλλουμε μια καλή πρόταση για την ηλεκτρονική κάρτα παροχής υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρεμπέσιους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Είπαμε ότι αυτή η κάρτα είναι αμφιλεγόμενη η Κομισιόν πιστεύει ότι η παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά θα διευκολυνθεί. Ε, όμως ε, δεν ισχύει αυτό αφού ήδη υπάρχει σύστημα αναγνώρισης των επαγγελμάτων. Η ηλεκτρονική κάρτα λοιπόν εδώ είναι διπλή δουλειά. Στη Γερμανία, τη χώρα μου, η επαγγελματική κατάρτιση είναι αποκεντρωμένη. στην Γερμανία ε, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα αναγνώρισης λοιπόν. Επίσης θα υπάρξει πρόβλημα για να εξευρεθούν οι ομόλογοι για να συνεννοηθούν κάθε φορά. Μια κεντρική λοιπόν διοίκηση ε, θα ε, υπονόμευε το σύστημα της Γερμανίας, το οποίο είναι αποκεντρωτικό. Δεν βλέπω λοιπόν ειδικά για τη χώρα μου κανένα όφελος. Επίσης υπάρχει ο φόβος ότι μέσα από την κάρτα αυτή ε, η ισοτιμία των ε, τίτλων σπουδών ε, επιβάλλεται άνωθεν. Εμείς δεν θέλουμε ισοτιμία πιστοποιητικών εκπαίδευσης άνωθεν επιβεβλημένη, διότι έτσι υπονομεύεται ο δίκαιος ανταγωνισμός. Επίσης, οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 156 της ε, ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης το απαγορεύουν αυτό. Ε, η επιβολή επίσης των ισοτιμία της ισοτιμίας προσκρούν και σε άλλες παραμέτρους που αφορούν και το θέμα της ασφάλισης με διαφορετική ποιότητα ε, των διπλωμάτων εκπαίδευσης ε, μπορεί να υπάρξουν διαφορές. Η υποχρέωση λοιπόν ασφάλισης ε, αλλοδαπών εργαζομένων θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Ορισμένες προτάσεις εδώ δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Θα πρέπει να μπορούμε να δεχόμαστε και την λειτουργία της αγοράς. Συμφωνώ ε, και με τους προηγούμενους ομιλητές ότι ε, παραβιάζεται η αρχή της ε, αναλογικότητας και της ρύθμισης για την ασφάλιση. Κάποια προτάσεις είναι παράλογες, οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι σε αυτή τη φάση να απορρίψουμε το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Ρίνα Ρόνια Κάρη. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι αναφερθήκατε στα θέματα που τονίσαμε μέσα από τις τροπολογίες, ε, δικαιολογήσατε την ε, απόρριψη ε, και συμφωνώ μαζί σας. Πολλοί πολίτες ε, έχουν πρόβλημα με το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πολλοί λένε ότι οι εταιρείε χρησιμοποιούν την ενιαία αγορά για να πηγαίνουν πέρα δόθε τους εργαζομένους και να τους ε, πιέζουν. Αυτό θα διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο για τις εταιρείε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι βεβαίως θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα κάνει ελέγχους η χώρα ελέγχου και θα, η χώρα υποδοχής ε, και θα εξασφαλίζει σωστές συνθήκες. Ποιος όμως ε, έχει τον έλεγχο των συνθήκων που πρέπει να ισχύουν. Είναι προφανές ότι πρέπει να απορρίψουμε ολόκληρη την πρόταση. Δεν υπάρχει λόγος να ε, επιχειρούμε εμβαλωματικές προτάσεις. Και κατόπιν τούτου είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις δυνατότητες ε, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, θα βγάλουμε τον κατασκευαστικό τομέα, θα, η χώρα υποδοχής θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες, ε, δεν θα υπάρχει δυνατότητα η Κομισιόν να κάνει εκτελεστικές πράξεις και διατάξεις και να δούμε προσεκτικά πώς λειτουργεί σήμερα το σύστημα τι αδυναμίες έχει, πώς μπορεί να αξιοποιήσει ε, τα δεδομένα αν δεν είναι ενημερωμένο. Ε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα IMI, ε, το σύστημα πληροφόρηση για την εσωτερική αγορά. Είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ιδέα πίσω από την πρόταση της Κομισιόν, κατά τη γνώμη μας, ε, είναι λογική. Πρέπει να διευκολύνουμε τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Αλλά οι αδυναμίες είναι πολλές στην πρόταση της Κομισιόν. Οπότε το θέμα που τίθεται είναι θα την απορρίψουμε συνολικά ή θα προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε. Η θέση μας είναι ότι προτιμούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ε, επαναδιατυπώσει την πρόταση. Αυτό θα ήταν η πρώτη επιλογή. και οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι. Παρ' όλα αυτά όμως καταθέσαμε τροπολογίες για να ε, καταδείξουμε τις αδυναμίες. Μέσα από την κατάθεση τροπολογιών αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να αναδείξουμε τις αδυναμίες. Πιστεύουμε πρώτον ότι η κάρτα δεν μπορεί να είναι αορίστου χρόνου. Πρέπει να έχει ημερομηνία λήξεως Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για να ελέγχουμε την ορθότητα των πληροφοριών, η προστασία των πελατών και χρηστών υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής ε, δεν παρουσιάζεται πολύ καλά στην πρόταση. Άρα και εδώ χρειάζεται περισσότερη εργασία, όπως και η υποχρεωτική ασφάλιση και υπάρχουν και κάποιες άλλες αδυναμίες που αναφέρονται στις τροπολογίες μας. Αυτή είναι η θέση μας που είναι λίγο περίπλοκη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι. Ευχαριστώ. Είναι κανείς άλλος από την ε, ομάδα FTD. Ο κύριος Μαρτάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να προσθέσει κανείς βέβαια τα κοινωνιστικά εμπόδια με τη θέσπιση αυτής της ηλεκτρονικής κάρτας ευρωπαϊκών υπηρεσιών φαίνεται εκ πρώτης ότι είναι μια καλή ιδέα, μια καλή λύση. Δυστυχώς όμως εδώ έχουμε ως στόχο να καταπολεμήσουμε τη θέσπιση φραγμών όσον αφορά τις διασυνορικές υπηρεσίες. Δηλαδή, το κείμενο περιορίζει την αρμοδιότητα ή τη δικαιοδοσία των κυρίαρχων κρατών για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην επικρατεία τους. Επίσης, βλέπουμε να υπάρχει το φαινόμενο ψευδών αυτοαπασχολουμένων, το οποίο υπόθηκε, και να έχουμε επίση τεχνητές μορφές απόσπασης. Έχουμε το κοινωνικό dumping, το οποίο επιτρέπει στους ξένους να μην χρειάζεται να ακολουθήσουν διάφορες διαδικασίες όσον αφορά διοικητικές διαδικασίες όπως οι Η συγγήτρια, η οποία σε χαίρο για τη δουλειά με εκπλήσει μάλιστα, γιατί εκφράζει τον σκεπτικισμό της, αλλά ότι είναι υπέρ των θέσεων της στην ε, γνωμοδότηση. Παρόλο που έχουμε κάποια τεκμηριωμένη γνωμοδότηση από ένα Εθνικό Κοινοβούλιο, το Αυστριακό Κοινοβούλιο, έχουμε το Γερμανικό Κοινοβούλιο, έχουμε και το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τα οποία μας προειδοποιούν σε σχέση με την εφαρμογή ή όχι αυτής της οδηγίας. Και καταλήγοντας, να σας πω ότι δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την Άγνες για, από τους σοσιαλιστές δηλαδή η μοναδική λύση είναι η παραπομπή του κειμένου στην ε, Κομισιόν και η Κομισιόν να δουλέψει κάπως περισσότερο και να μας υποβάλει, να μας παρουσιάσει κάτι το οποίο θα είναι εφικτό. Αυτό προτείνω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, then Ευχαριστώ. Θα δώσω λόγο Σαντέ. Παρακαλώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου σε σχέση με την πρόταση της ε, Κομισιόν γιατί χρειάζεται πολύ δουλειά πραγματικά αν θέλουμε όντως να προωθήσουμε το κείμενο αυτό. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία εκ μέρους των επαγγελματιών μας ιδιαίτερα των Γάλλων να αναφέρω κάποια προβληματικά ζητήματα που ανέφεραν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Το πρώτο βεβαίως αφορά την αρχή της ε, αυτόματης έγκρισης, κάτι το οποίο απειλεί να επαναεισαγάγει την αρχή της χώρας προέλευσης και το οποίο μας ενσυχεί. Άλλο ένα θέμα προβληματικό είναι η διορία δύο εβδομάδων που έχουν στην διάθεσή τους οι χώρες μέλη για να απαντήσουν. Και αυτό βεβαίως χωρίς να διαθέτουν πραγματικά ουσιώδη δηλαδή αυτά έγγραφα. Νομίζω ότι βεβαίω θα πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτά τα θέματα και να παραθέσω και το θέμα της διάρκειας, της ε, επαορίστων διάρκειας της κάρτας αυτής. Εγώ νομίζω θα πρέπει εδώ να θεσπίσουμε μια χρονική διάρκεια ισχύω της κάρτας, αλλά επίσης και την δυνατότητα αναθεώρησης των πληροφοριών όσον αφορά την παροχή της κάρτας αυτής. Άλλο ένα πρόβλημα είναι το ότι η αρχή της κάρτας, η διαχείριση της βασίζεται σε κάποια περίπλοκα ζητήματα και σε ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία φαίνεται να μην είναι κατάλληλα και από τα οποία από ό,τι φαίνεται λείπει κάποια σύγχρονη και επίκαιρη λειτουργικότητα αποτελεσματική και προσβάσιμη σε όλους. Και τέλος ένα τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η εφαρμογή αυτής της ηλεκτρονικής κάρτας νομίζω ότι θέτει κάποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την διάρθρωσή της, που φαίνεται να είναι κάτι το δυσχερές σε σχέση με άλλες υπάρχουσες διατάξεις, όπως τα νέα κέντρα εξυπηρέτησης τα οποία προβλέπονται από την οδηγία, ή αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, που ανέκυψε από την οδηγία για τα προσόντα, τα επαγγελματικά. Αυτά από εμένα και νομίζω ότι πραγματικά οι εισηγητέ μα έχουν τεράστια δουλειά μπροστά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σόιντροβα. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτή η πρόταση οδηγίας απέβλεπε στο να τηρήσει μακροχρόνιες ε, στοχεύσεις όσον αφορά το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς. Εμείς ελπίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε άρει όλους τους φραγμούς στην κυκλοφορία ατόμων και αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Η συζήτηση όμως εδώ στην Επιτροπή μας δείχνει ακριβώς ότι αυτό δεν ισχύει και δείχνει μάλιστα ότι οι χώρες μέλη αυτή τη στιγμή φοβούνται το κοινωνικό dumping και ανησυχούν για θέματα όπως ε, τι ισχύει με την ε, σχέση νομοθεσία σε συγκεκριμένε χώρες, ιδιαίτερα σε χώρες προέλευσης. Οπότε, ε, με επιτρέψαμε να πω ότι εδώ με κάποιο τρόπο δημιουργούμε προστατευτικά μέτρα, μέτρα προστατευτισμού. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να προτείνει ένα εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει την κυκλοφορία των υπηρεσιών. Βεβαίως, φαντάζομαι ότι δεν ήταν στόχος της Κομισιόν να διευκολύνει την παραβίαση της νομοθεσίας των χωρών μελών. Όμως η κατάσταση στις χώρες μέλη είναι αυτή που είναι σήμερα. Καταλαβαίνω αυτούς που έχουν συγκεκριμένε θέσει και βλέπω ότι είναι δύσκολο το Κοινοβούλιο να επιστρέψει την οδηγία στην Κομισιόν επειδή εμείς ε, θα λέει κανείς ότι δεν θέλουμε να άρουμε τους ε, φραγμούς θα μας έλεγε και θα μας κατηγορούσε ότι δεν θέλουμε να άρουμε τους φραγμούς αλλά εμείς θα πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα τεχνικό μέτρο και να σας πω ότι στην αρχή θεωρούσα ότι ως μέτρο αυτό είναι αρκετά προβληματικό αλλά καταλαβαίνω τελικά ότι συμμορφώνεται με το πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Αν έχουμε λοιπόν τελικά μια ηλεκτρονική κάρτα και ένα αντίστοιχο κανονισμό, αυτά θα πρέπει να είναι ε, συμμορφωμένα με αυτά που προβλέπει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Χάκεν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ συναδελφοί. Νομίζω ότι κατά διάρκεια της συζήτηση έγινε σαφέστερο ποιες είναι οι θέσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Είναι σαφές και από τις ε, τροπολογίες, γκούες, σοσιαλιστές και νομίζω ότι αυτό μπορώ να πω τώρα ότι θα καθίσουμε τους και όλους να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και στην συνάντηση των σχεδόν εισηγητών θα το αποφασίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 22 και 23 του Γενάρη του χρόνου. Και στην ΕΚΟ 21-22 και θα πάμε στο, το Μάρτι στην Ολομέλεια. Πάμε στο σημείο 9 της ημερησίας. το νομοθετικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής κάρτας, δηλαδή το ίδιο θέμα από διαφορετική οπτική σκοπιά. Κυρία Σοντερόβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Δεν θέλω να επαναλάβω τη συζήτηση που είχαμε τη γενικότερη. Πρέπει όμως να υπενθυμίσω ότι αυτή η, ηλεκτρονική, η Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Κάρτα Υπηρεσιών αποβλέπει στην ευκόλυση της παροχής υπηρεσιών και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τελικός στόχος αυτής της ε, πρώτας οδηγίας. Σύμφωνα όμως με τις τροπολογίες σας βλέπω ότι ανησυχείτε ότι στην ουσία υποβαθμίζει τις αρμοδιότητες των χρόνων μελών και το καταλαβαίνω. Η ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών αποβλέπει στην λαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου αυτό καταλαβαίνω εγώ, αλλά καταλαβαίνω και πάλι τις ανησυχίες σας. Οι υποποθέσεις παροχής αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει βεβαίω να είναι σύμφωνες με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία των χωρών μελών. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαι τελείω αντίθετη με την τροπολογία που προτείνει την ε, καταψήφιση αυτής τη πρόταση. Έχουμε 204 τροπολογίε που κατατέθηκαν ποικίλη φύση. αλλά μπορούμε να πούμε ότι επικεντρώνονται στα εξή. Καταρχά, η σιωπηλή αποδοχή που εγκρίνει την ισχύ της ηλεκτρονικής κάρτας και η διασφάλιση των αρμοδιοτήτων των χωρών μελών αφορά την επέκταση της κάρτας και της καθυστερήσεις. Μετά. Η κάρτα και η κατεξοσοδότηση νομοθετικής πράξης της Κομισιόν. Αυτά είναι τα κυριότερα πεδία. Θα έχουμε βέβαια και συμβαστικές προτάσεις τροπολογίας που θα λάβουν υπόψη τις ανησυχίες σας. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν βεβαίως και νομικές προβλέψεις που απορρέουν από τις γνωμοδοτήσεις που κάποιοι από εσά θα ήθελαν να καταργήσουν όσον αφορά την παροχή και την ε, επέκταση αυτών των υπηρεσιών. Πάντως η τωρινή οδηγία υπηρεσιών για την ενιαία αγορά επιβάλλει τον κανόνα της σιωπηλή αποδοχής όσον αφορά τις ε, εγκρίσει των διαδικασιών αδειοδότηση. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να διατηρηθεί. Παρομοίω, η ίδια οδηγία προβλέπει ότι οι εγκρίσεις μπορεί να περιορίζονται χρονικά μόνο εάν ανανεώνονται αυτομάτως. Κάποιοι από εσά προτείνατε σχετικά κάποια όρια. Είναι όμως σημαντικό αυτά τα όρια να συνδυάζονται με την ε, ρήτρα της αυτόματης ανανέωσης. Θα ήθελα να σας καλέσω να λάβετε υπόψη σας άλλη μια εναλλακτική λύση ως προσέγγιση από τη στιγμή που η βιομηχανία της οικοδομής είναι κάθετα αντίθετη με αυτή την κάρτα και θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τις υπηρεσίε προς επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι η υπηρεσία αυτής της μορφής με την ηλεκτρονική κάρτα είναι εθελοντικής μορφής. Δηλαδή θα πρέπει να αποτελεί μια εναλλακτική λύση όταν εισέρχεται κάποιος στην αγορά κάποιας χαράς, χώρας μέλου, μέλους. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες να έχουν εγγυήσει. Θα πρέπει να τα έχουμε λοιπόν όλα αυτά κατά νου όταν θα συζητήσουμε τις τροπολογίες μας και ανάλογα με την λειτουργικότητα και την επιτυχία της κάρτας αυτής θα μπορούσαμε μελλοντικά ενδεχομένως να διευρύνουμε το πεδίο της κάρτας αυτής και στον τομέα της οικοδομής και νομίζω θα ήταν αρκετά σωστό να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να περιορίσουμε το πεδίο αλλά θα πρέπει να είμαστε και ελαστικοί γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μην θέσουμε σε κίνδυνο όλη την πρόταση και τις δυνατότητές της. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε ένα κοινό έδαφος εδώ και συμβασμούς, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για να το κάνουμε αυτό. Οπότε προσλέπω στη συζήτηση που θα κάνουμε και ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, κυρία Σόιντρομα η κυρία Γιουγκέριος από τους σοσιαλιστές. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπα στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και για αυτό το σημείο, αυτά που είπα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ, η κυρία Τρεμπέζιος. Η κυρία Γιουγκέριος νομίζω πολύ σωστά είπε ότι επί της ουσίας συζητήσαμε το θέμα. Η συγγήτρια έχει κάποιες νέες προτάσεις, σημεία. Όμως δεν θα βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση με αυτές τις νέες προτάσεις. Δημιουργούμε μια νέα δομή και ουσιαστικά δεν αντιστοιχεί στην δομή της δικής μας χώρας τουλάχιστον. Πολύ συγκεντρωτική δομή. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή εκφραστήκαμε στο προηγούμενο σημείο, η δική μας θέση είναι κοινή και για τις δύο αυτές ε, προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος, κυρία Άρντεν. Και εγώ Πραγματικά δεν έχω να προσθέσω πολλά σε σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως. Όπως είπε η συγγήτρια, σκοπός είναι να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό είναι ο σκοπός. Δεν νομίζω όμως ότι με αυτές τις προτάσεις θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο και η τροποποίηση αυτής της πρότασης ε, είναι τόσο από όλε τις πλευρές και σημαντική που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία όπως η κυρία Γκάριν εξάλλου νομίζω ότι υπάρχουν και θέματα θέμη του ανταγωνισμού για τους αυτοαπασχολούμενους κτλ. κτλ. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόταση αυτή δεν είναι σωστά διαρθρωμένη και Βεβαίως όπως θα συζητήσουμε και στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, δεν ξέρουμε αν μπορεί να τροποποιηθεί. Από τη μία μας λένε ότι είμαστε υπέρ του προστατευτισμού. Από την άλλη, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν απάτες, ότι το σύστημα δεν λειτουργεί και ότι η πρόταση αυτή η καινούρια δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά αυτές τις αδυναμίες, τότε και αυτό ισχύει για πολλά συστήματα, για πολλές πτυχές του συστήματος αυτούς. Δεν είμαι ειδική, αλλά από ό,τι διάβασα δεν αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα με αυτήν εδώ την πρόταση. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί και σαν πολιτική ομάδα θεωρούμε ότι δεν ε, μπορούμε να στηρίξουμε προς το παρόν τουλάχιστον αυτές τις προτάσεις. Αλλά παρόλα αυτά περιμένω να δω τι θα γίνει στην συνάντηση των σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτά που είπα στο προηγούμενο σημείο θεωρώ ότι ισχύουν και εδώ και γι' αυτό και θα πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω προς την εισηγήτρια και τα εισαγωγικά της σχόλια. Είναι το σύστημα αυτό προαιρετικό και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το στηρίξουμε. Από την άλλη, αυτό το προαιρετικό ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να πούνε ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν αν ναι ή όχι θα συμμετέχουν στο σύστημα. Και με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται ότι ο κατασκευαστικός τομέας εάν απορρίπτει το σύστημα αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε εμείς να το δεχτούμε. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι προς το παρόν αποκλείεται ο κατασκευαστικός τομέας και θα ενσωματωθεί αργότερα. Αυτό και μόνο δείχνει για ποιο λόγο πρέπει να απορρίψουμε όλη την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζανότκα. Ναι. Ένα έχω να προσθέσω. Ένα μόνο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια καταρχήν. Την εισηγήτρια την Ατίνα Σόντροβα. Πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα και, και εγώ προσβλέπω στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να δούμε αν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ε, θέσεις μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Μάτα, ο κύριος Μάτα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα κι εγώ. Από το σημείο που πιστεύουμε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Κάρτα Υπηρεσιών δεν είναι κάτι που μπορούμε να στηρίξουμε. Ας αφήσουμε τις ε, νομικές πτυχές γιατί χάνουμε το χρόνο μας πραγματικά αν το συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα το γνωρίζετε. 26 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή και το Μάρτιο στην επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή. Όσον αφορά την Ολομέλεια δεν έχουμε ακόμα τις ημερομηνίες. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας. Όπως ξέρετε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει η πρωτοβουλία για την οργάνωση της Αφρικανικής Εβδομάδας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που απορρέει από την συνάντηση κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης που θα λάβει χώρα στο Αμπιτζάν πολύ σύντομα. Θέλουμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας, γι' αυτό και έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονες από την Αφρικανική Ήπειρο Εμείς σαν ε, Επιτροπή Απασχόλησης θα επικεντρωθούμε στα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας Θα μιλήσουμε για τις θέσεις απασχόλησης και για τις μελλοντικές προοπτικές ε, ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων. Uh, Εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, συνήθως επικεντρωνόμαστε σε θέματα ανεργίας, μελλοντικών προοπτικών της αγοράς απασχόλησης, απασχόληση προοπτικές για τους νέους, το θέμα της Αφρικής είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονες, άτομα που μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο για τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σας παρακαλώ μπορείτε να πάρετε το λόγο, να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση ποιος είστε. Και βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των νέων γενιών και των νέων. Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορείτε να είστε όρθιοι και να συζητάτε μέσα στην αίθουσα. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Good morning. Um... Καλημέρα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, μου είπα να παρουσιαστώ. Είμαι η Σύνθια Σάμουελ Ολόντζουβον. δύσκολο όνομα να το προφέρομαι. Εργάζομαι για την ε, Αφρική ε, στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και είμαι επικεφαλής της, του Τμήματος Προγραμματισμού για την Αφρική. Καλημέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Είμαι ο Λου Κρίστιανσεν. Ε, είμαι στην Παγκόσμια Τράπεζα υπεύθυνος για τα οικονομικά της περιφέρειας της Αφρικής. Κουτσιλάη, Παγκόσμια Τράπεζα, ε, στον τομέα των συμπράξεων. Δεν είμαι όμως ομιλητής σήμερα. Ο συνάδελφος μου Μάθιου ε, είναι στις Βρυξέλλες και εξαιρετικός στην ε, όλη διαδικασία η οποία με έφερε εδώ μου είπα να μιλήσω για επενδύσεις στους νέους στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του πέμπτου διαλόγου Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχει τη μορφή ε, συνόδου κορυφής. Θα παρουσιάσω ορισμένα θέματα μέσα από το πρίσμα της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να έρθουμε σε αυτήν τη σημαντική συζήτηση που δεν είναι σημαντική μόνο για την Αφρική και την Ευρώπη αλλά έχει παγκόσμια σημασία. Η παρέμβασή μου θα μπει σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο ζήτημα που αφορά τη συζήτηση αυτή είναι ότι το 2045 εκτιμάται ότι 50% των νέων της Αφρικής θα είναι Αφρικανοί μέχρι το 2045. Εκτιμάται επίσης ότι το 2, μέχρι το 2040 η αγορά εργασίας στην Αφρική θα είναι πολύ σημαντική αριθμητικά. Στα πλαίσια της έκθεσης για τους νέους το 2017 που εκδόθηκε χθες, ε, αναφέρεται ότι αν συγκρίνουμε με το 2009, παγκόσμια βελτιώθηκε η κατάσταση απασχόλησης των νέων, αλλά ακόμα η κατάσταση είναι απέχει από το να είναι ικανοποιητική, ιδιαίτερα αν δούμε την ποιότητα των θέσεων εργασίας στην Αφρική σε κάποιες χώρες. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω επιτάπητος για να το συζητήσουμε είναι μία από τις αρχές της διακήρυξης της Φιλαδέλφια του 1945 της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που λέει ότι η φτώχεια οπουδήποτε αποτελεί απειλή για την ε, ευημερία οπουδήποτε είτε είναι σε εθνικό επίπεδο η φτώχεια είτε είναι σε υπηρετικό επίπεδο ή αν είναι σε επίπεδο παγκόσμιο Όλα αυτά λοιπόν αν τα συνδυάσουμε βλέπουμε ότι υπάρχει αδύρυτη ανάγκη να ε, καταπιαστούμε σοβαρά με το θέμα της απασχόλησης των νέων στην Αφρική και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Ε, πολύ σοβαρά. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται μόνο για ένα θέμα ε, εξωτερικό που δεν μας αφορά. Είναι βασικό θέμα αν δούμε το μέλλον της εργασίας και αν δούμε ποια θα είναι η εικόνα της αγοράς εργασίας στο μέλλον. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Εις ό,τι αφορά τα μέσα, τους τρόπους για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό ε, των νέων αυτών που, που έχουν σημασία δημογραφική και τώρα και στο μέλλον ε, το ψήφισμα του 2012 ε, που, για την εργασία των νέων μας δίνει μια καλή βάση. Θα ήθελα να υπησέλθω σε κάποια θέματα που πρέπει να δούμε πολύ πιο προσεκτικά. Πρώτον, η ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται σε πολλές θέσεις εργασίας. Πολλές φορές δίνεται έμφαση στην πρόθεση της ανάπτυξης. Πολύ ωραία. Αλλά αν δεν υπάρχει και άφθονη απασχόληση, δεν θα έχουμε ανάπτυξη, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της φτώχειας. Μια, ένα βασικό θέμα σε όλα αυτά είναι να διασφαλίσουμε ότι οι θέσεις εργασίας, κυρίως για τους νέους αξιοπρεπή δουλειά, Ε, ε, συμπεριλαμβάνονται και στη δημοσιονομική πολιτική. Ανάπτυξη λοιπόν, ανάπτυξη αλλά και θέσεις εργασίας. Δεύτερο θέμα. Πρέπει να εντοπίσουμε τους βασικούς τομείς που είναι εντατικοί από άποψη απασχόλησης, ιδιαίτερα απασχόλησης των νέων. Και να δούμε τι αδυναμίες υπάρχουν, ε, τι είναι οι παράγοντες απόθεσης για τους νέους. Θα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι τομείς, θα πρέπει να δούμε ε, τρόπους να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε νέα ταλέντα. Η γεωργία είναι ένας τομέας σημαντικός, ο κατασκευαστικός τομέας και κάποιοι άλλοι που θα αναφέρω αργότερα. Ένας τρίτος τομέας αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων, ώστε να είναι απασχολησίμοι δεξιότητες μέσα από εκπαίδευση, κατάρτιση, διάφορες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Αργότερα θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη συζήτηση. Ένας τέταρτος βασικός τομέας αφορά τα δεδομένα και την προώθηση της, ε, των υπηρεσιών απασχόλησης. Στην Αφρική, μια πρόκληση που έχει εντοπιστεί και αυτό φάνηκε καθαρά, είναι το θέμα των δεδομένων. Για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε ε, τις προοπτικές αξιοπρεπούς απασχόλησης πρέπει να επενδύσουμε στην ε, πληροφορία, σε συστήματα πληροφοριακά για την αγορά εργασίας, να έχουμε πληροφορίες που θα, χαράξουν, που θα βοηθήσουν να χαράξουμε πολιτική και να την ε, εφαρμόσουμε μετά. Υπάρχουν τρεις άλλοι τομείς που θα ήθελα να προσέξουμε περισσότερο. Πρώτον, η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξή της. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί κάθε νέος να γίνει επιχειρηματίας, αλλά αυτοί που μπορούν να γίνουν θα πρέπει να υποστηριχθούν για να γίνουν καινοτόμοι, να παραγωγικοί ε, μέσα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Και εδώ χρειάζονται επενδύσεις. Ε, πόροι, οικονομικοί και άλλοι, για να προαχθεί η επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει μία λύση για όλες τις καταστάσεις. Ιδιαίτερα στην Αφρική Υπάρχουν πολλές ευαλωτότητες και εύθραυστες καταστάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι τρόποι παρεμβάσεων σε αυτά τα δεδομένα πρέπει λοιπόν να ε, προσέχονται ιδιαίτερα. Σε επίπεδο Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ΑΕΛΟ στην Αφρική έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να λάβουμε υπόψη μας τις τροτότητες αυτές. Αυτό έγινε το 2015. Το Ιούνιο του 2017 σε παγκόσμιο επίπεδο η Διεθνής ε, Διάσκεψη Εργασίας ε, νέκρινε συστάσεις σε όλους αυτούς τους τομείς για την προώθηση αξιοπρεπούς απασχόλησης ε, και ε, πάνω στη βάση της ειρήνης και της ανθεκτικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να Προαχγεται η αποσχολησιμότητα των νέων ε, ακόμα και σε έθραυστες καταστάσεις. Εδώ έχουν γίνει πολλά. Τέλος, οι συμπράξεις, πολύ σημαντικό θέμα, οι εταιρικέ σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε περιφερειακό, σε εθνικό επίπεδο. κανένας φορέας δεν μπορεί να απασχοληθεί και να λύσει το θέμα της απασχόλησης των νέων μόνος του. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όλοι για αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Υπάρχει ένα ε, σχετικό ε, πλαίσιο για την υποστήριξη των κρατών μελών ε, ώστε να διατυπώσουν μια σαφή απάντηση, αντίδραση ε, στις ανάγκες απασχόλησης των νέων στις χώρες τους. Αυτή η πρωτοβουλία ε, είναι μια πλατφόρμα που βοηθάει τις χώρες να ε, λειτουργούν ως DG8 και DG4. έχουμε ε, διατυπώσει μια πολιτική στην ILO για να προχωρήσουμε μαζί και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των νέων λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές τάσεις και τις μελλοντικές προσδοκίες ε, ε, από την αγορά εργασίας. Σταματώ εδώ και θα επανέλθω κατά τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κρίστιανσες από την Παγκόσμια Τράπεζα για μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Μια στατιστική που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι μέχρι το 2050 αναμένουμε να έχουμε 2 δισεκατομμύρια πληθυσμό στην Αφρική και 700 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Αυτό μας δείχνει ακριβώς τον μελλοντικό ρόλο της Αφρικής, το άμεσο σχετικά μέλλον. Ξέρουμε τα γραφήματα αυτά σε σχέση με τον πληθυσμό και μας δείχνουν δηλαδή ότι η πυραμίδα του πληθυσμού αριστερά για την Αφρική βλέπετε ότι αποτελεί ένα τρίγωνο στο σκελές, δηλαδή έχουμε πολλά εκατομμύρια νέων ανθρώπων και κυρίως νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει την δομή την πληθυσμιακή της Αφρικής. Οπότε δεν έχουμε μόνο πολλούς νέους, αλλά έχουμε πολύ περισσότερους. Είχαμε κάποια οικονομική ανάπτυξη, κάποια ανοίγματα, έχουμε κάποιες φιλοδοξίες και προσδοκίες που μεγαλώνουν, αλλά έχουμε και πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και ένας από τους ε, σημαντικούς ε, δείκτες μας μας το επιβεβαιώνει αυτό όσον αφορά δηλαδή την εκπαίδευση και αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την απασχόληση για αυτή την νεολαία. Εκεί λοιπόν που βλέπουμε ευκαιρίες στην Αφρική αυτή τη στιγμή πολλοί απασχολούνται στην γεωργία το δεξί γράφημα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις επίσης στην άτυπη εργασία έχουμε μεγάλη μορφή απασχόληση. Δηλαδή φαίνεται ότι στον επίσημο τομέα δεν δημιουργούνται αρκετές θέσεις γι' αυτό έχουμε ισχυρή παρουσία της άτυπης εργασίας. Όπως υπόθηκε λοιπόν και προηγουμένως, είχαμε διάφορα προγράμματα, πολλά προγράμματα που ισχύουν και καιρό. Και τα περισσότερα από αυτά για την απασχόληση των νέων κάνουν παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση των προσόντων τους για τις επιχειρήσεις, για την καθημερινότητά τους, για την πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση. Υπάρχουν όμως πολλές μελέτες που εξετάζουν αξιολογήσει αυτών των προγραμμάτων και δείχνουν ότι ο αντίκτυπός τους ήταν χαμηλός. 20% είχαν θετικό αντίκτυπο και στατιστικά φαίνεται ότι αυτός ο αντίκτυπος δεν είχε τόσο μεγάλη στατιστική απήχηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να σας απασχολήσει να σκεφτούμε δηλαδή το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Προγράμματα λοιπόν απασχόληση των νέων στο παρελθόν επικεντρώνονταν, επικεντρώνονταν κυρίως στην πλευρά της, της παροχής, δηλαδή προσόντα όσον αφορά το, το ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά θα πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό. Και πάλι λοιπόν, μετά από αυτά που είπε η προλαλήσασαν, να σας πω ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα και αποτελεί ένα θέμα εταιρική σχέσης που ήδη υπάρχει από το 2014. Δηλαδή, εδώ έχουμε το δημόσιο τομέα, βλέπετε τους ε, εταίρους από το ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών υπάρχουν εταίροι, ώστε να δοκιμάσουμε και να αναζητήσουμε πιλωτικές λύσεις που θα έχουν καταλητικό αποτέλεσμα, όχι για άμεση επιτυχία, αλλά να έχουν καταλητικό μελλοντικό ρόλο. Αυτοί είναι κάποιοι από τους εταίρους. Όπως βλέπετε έχουμε κάποιους σημαντικούς φορείς από το ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και κυβερνήσεις. Έχουμε λοιπόν και πρόγραμμα για τους νέους στα πλαίσια της Παγκόσμιας Τράπεζας που ακολουθήσαμε για 15 χρόνια. Και εδώ έχουμε λοιπόν άλλη μια εταιρική σχέση που προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Νομίζω αυτό που είναι σημαντικό όταν μιλάμε για απασχόληση είναι βεβαίως το να έχει κανείς μια δουλειά και η ποιότητα της δουλειάς, της θέσης εργασίας. Νομίζω το κυριότερο προσπαθεί να κάνει αυτή η εταιρική σχέση και αυτό που είναι νέο είναι όχι μόνο το να επικεντρωθούμε στην πλευρά της προσφοράς, δηλαδή στην παροχή δεξιοτήτων, ε, εκπαίδευση δηλαδή εν εισόδου στην αγορά, αλλά προσπαθούμε να εργαστούμε και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα, μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Προσπαθούμε δηλαδή να αναπτύξουμε την αλυσίδα αξίας, εξετάζοντας τους περιορισμούς για τις δύο πλευρές. Όσον αφορά τη ζήτηση, βεβαίως μιλάμε για την ε, ανάπτυξη που φέρνει η θέση εργασία και αφορά το ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως και για την ανάπτυξη του δημοσίου τομέα χρειάζονται πολλέ μακροοικονομικές ε, πολιτικέ σταθερότητε, σταθερότητες κτλ. Αλλά αυτό είναι κάπω εκτό ε, πεδίου βεβαίω αυτών των προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων. Αλλά μπορούμε να κάνουμε αρκετά εδώ. Για κάποιου τομεί έχουμε περισσότερη ένταση εργασία σε σχέση με κάποιου άλλου τομεί. Μπορούμε λοιπόν να το διευρύνουμε αυτό. Α πούμε, για τη γεωργία χρειαζόμαστε πρόσβαση στι αγορέ δεν είναι αυτό ο σκοπό η γεωργική παραγωγή, είναι παραγωγή για πρόσβαση στι αγορές. Οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, να αναπτύξουμε ενδεχομένω την αγορά και ενισχύοντα του γεωργού ώστε να παράξουν για αυτέ τι αγορέ με έναν τρόπο ολοκληρωμένο. Στην ουσία, εξετάζουμε τι παρεμβάσει τι ανθρώπινε και επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσπαθώντα να καλύψουμε κενά πληροφόρηση όπου υπάρχουν. Εξετάζουμε ε, πεδία όπου πραγματικά υπάρχει ε, δυνατότητα για ανάπτυξη της αξίας. Έχουμε δυνατότητα λοιπόν αύξησης παραγωγής, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα γι' αυτό, για αύξηση της παραγωγής από τους ε, γεωργούς. Οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε με διάφορους εταίρους ταυτόχρονα, ώστε να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση. Και αυτό ήταν ένα και μόνο παράδειγμα σας έδωσα στα πλαίσια Οπότε το πρόγραμμα αυτό έχει αυτή την εταιρική σχέση που βρίσκεται στη δεύτερη φάση. Και έχουμε δύο κύριους τομείς, καινοτομία και εκπαίδευση κατάρτιση. Στην καινοτομία θέλουμε να αναπτύξουμε πιλωτικά μια και πάλι ολοκληρωμένη προσέγγιση, εξετάζοντας βέβαια και τις δύο πλευρές και τις προσφοράς και τις ζήτησης. Κάνοντας αυτό, ελπίζουμε να πετύχουμε συνέργειες ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη, ένα πιο πλήρες αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας αλυσίδας για να ξεπεράσουμε ας πούμε προβλήματα συντονισμού. Μπορεί να γίνει και μέσω χωρικής ανάπτυξης όπου θα έχουμε ας πούμε, την υλοποίηση μιας ολοκλήρωσης σε διάφορους τομείς. Αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να, ξέρετε, να προσεγγίσουμε και να πετύχουμε την ολοκλήρωση. Στο πρόγραμμα Υπάρχει μια διασύνδεση με το μελλοντικό φόρουμ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία για την Αφρική, για την απασχόληση των νέων στην Αφρική. Όπως ξέρετε, έχουμε πολλές συζητήσεις σήμερα για τις ψηφιακές δουλειές, ψηφιακές θέσεις εργασίας, η μικροεργασία, η... το freelancing και στον τομέα της ε, πληροφορικής. Βέβαια, υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό αλλά ταυτόχρονα αυτό απαιτεί οι ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν τη βάση τους και να ενισχύσουν την πρόσβαση στο ίντερνετ ας πούμε ώστε να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν ας πούμε πρόσβαση σε, στην κινητή τηλεφωνία εκτός από υποδομές όπως ηλεκτρικό ρεύμα κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε και τις βασικές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν για να ελοπίθουν όλα αυτά. Οπότε επικεντρωνόμαστε στα πλαίσια αυτού του προγράμματο στι ηλεκτρονικέ θέσει εργασία, στι ψηφιακέ. και κάνουμε μια αποτίμηση του τι ήδη γίνεται εδώ σε αυτό το τομέα και έχουμε συζητήσει με ενό οικονομολόγου στην Αφρική αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να υποβάλουμε μια έκθεση από την οποία θα πορεύουν διάφορε κατευθυντήριε γραμμέ σε σχέση με κάποια πιλωτικά προγράμματα. Αυτό, με δύο λόγια, είναι ο στόχος μας στα πλαίσια αυτής της εταιρικής σχέσης για την απασχόληση των νέων. Συνοψίζοντας, κάποια κύρια μηνύματα που θα θέλαμε να στείλουμε είναι ότι χρειάζεται μια ανάγκη, ότι, συγγνώμη, υπάρχει μια ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση, ότι θα πρέπει να έχουμε κατάρτιση βεβαίω για την αγορά, αλλά να δούμε το θέμα της κατάρτασης ε, γενικότερα εκεί όπου υπάρχουν κενά και αυτή η εταιρική σχέση ακριβώς αποτελεί ένα βήμα παραπέρα στο να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά και τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Ακούσαμε την πρώτη ομιλήτρια που είπε ότι είναι επίγον το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας στην Αφρική. Ο κύριος Κρίστενσεν, ο δεύτερος ομιλητής, είπε ότι βεβαίως πρέπει να κάνουμε και πολλά παραπάνω. Έχουμε και την κυρία Μοντέση από την Επιτροπή, η οποία εργάζεται με την Κεντρική και Δυτική Αφρική, κάνει τον συντονισμό της ανάπτυξης, αναπτυξιακής πολιτικής. Έχετε το λόγο. Θα μιλήσω γαλλικά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Η Σύνθια και ο Λίκ είπαν πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Όσον αφορά τη στρατηγική, την πολιτική που είναι ο τομέας της αρμοδιότητάς μου, θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία. Από το 2030, 400 450 εκατομμύρια νέοι θα φτάσουν στην αγορά εργασίας στην Αφρική, υπό Χασαχάρια και υπόλοιπη Αφρική και καθότι υπάρχει αυτή η σημαντική δημογραφική ανάπτυξη θα πρέπει να δημιουργούνται Εφτά ή 8 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες αυτών των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικές επί της οικονομίας και επί των ε, πολιτικών μας επαφών με την Αφρική. Οι νέοι, άνεργοι, απογοητευμένοι νιώθουν ε, ότι επικρατεί κοινωνική αδικία και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κοινωνικές εντάσεις, πολιτικές εντάσεις και ένα αίσθημα απογοήτευσης και ε, ενδεχομένως ε, δημιουργούν κίνητρα για να πλησιάσει κανείς ε, την τρομοκρατία και τη βία. Είναι λοιπόν κοινή η πρόκληση της Ευρώπης και της Αφρικής. Πρέπει να σκεφτούμε τους νέους, όχι μόνο τους νέους στην Ευρώπη, αλλά και τους νέους στην Αφρική, που είναι πολλοί, που ψάχνουν ε, ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Τι κάνουμε στην Ευρώπη. Και θα επικεντρωθώ κυρίως σε αυτό. Εδώ και χρόνια η προοπτική της βελτίωσης των ε, προοπτικών απασχόλησης για τους νέους είναι στο κέντρο της πολιτικής μας. Έχουμε μια κοινή προσέγγιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ένα κοινό έγγραφο που έχουμε υιοθετήσει εδώ και κάποιους μήνες που είναι ουσιαστικά η υλοποίηση της Ατζέντα 2030 με στόχους και την ανάγκη να βρούμε λύσεις στα προβλήματα της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες περιοχές, όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα παιδιά. Έχουμε καθορίσει προτεραιότητες, πρόσβαση στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση, τεχνική, επαγγελματική για όλους, μία προϋπόθεση για να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των νέων. Δεύτερος πρωταρχικός στόχος είναι να βρεθούν απαντήσεις και λύσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι εντοπισμός μιας αξιοπρεπούς εργασίας, ποιοτικής εργασίας για τους νέους αυτούς που θέλουν να βρουν νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές και νέες εταιρικέ σχέσεις. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα έχει διάφορες μορφές. Ο Λουκ μίλησε για την διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα διακυβέρνησης στις διάφορες αφρικανικές χώρες. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν χώρες πιο ασταθείς, άλλες περισσότερο ανεπτυγμένες. Σε όλες όμως αφρικανικές χώρες θα πρέπει να βελτιωθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της προσέλκυσης των επενδύσεων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι αυτές που κυρίως δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, των οποίων η ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί και να διευκολυνθεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα στα οποία στηρίζουμε την κατάρτιση. Παραδείγματο χάρη, όπω είπε ο Λουκ, την ε, εκπαίδευση γενικότερα, αλλά την επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση. Μεταξύ του 2014 και του 2020, πάνω από 1,5 δι έχει διατεθεί σε θέματα κατάρτισης και επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συν 200 εκατομμύρια για τις γενικότερες ε, πολιτικές συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης και άλλα 300 εκατομμύρια για το Erasmus Plus, ένα πρόγραμμα που νομίζω γνωρίζετε. Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη μέσω αυτών των κονδυλίων για τους νέους οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν δικές τους ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε και ο Λίκ, αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κατάρτισης και διακυβέρνησης. Διαθέτουμε κονδύλια για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, για τους νέους και ενίσχυση των δυνατοτήτων των εθνικών αρχών και κυβερνήσεων για να ενισχυθεί η δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης κυρίως σε κάποιους ε, τομείς που παρουσιάζουν περισσότερες ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Νίγηρας παραδείγματος χάρη ε, στον οποίο στηρίζουμε την κυβέρνηση στο νομοθετικό της έργο, στη διακυβέρνηση για την ε, στήριξη κάποιων τομέων στους οποίους μπορεί να δημιουργηθούν ε, θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Επίσης στηρίζουμε προγράμματα κατάρτισης για 6.000 νέους και βοηθούμε την ενσωμάτωση των νέων αυτών με μικροχρηματοδότηση, μικροπιστώσεις που δίνονται κατευθείαν στους νέους. Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για την στήριξη της σταθερότητας στην Αφρική και της αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Αυτό βεβαίως έχει από κοινού με τα ευρωπαϊκά προγράμματα προγραμματιστεί. Δίνουμε όμως συγκεκριμένη οικονομική στήριξη και τεχνική κατάρτιση στους νέους στην Αφρική. Αυτά είναι τα υπάρχοντα, τα ισχύοντα ε, προγράμματα. Για το μέλλον δημιουργούμε ένα νέο εργαλείο, ένα νέο σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων για την Αφρική με τρεις πυλώνες, χρηματοδότηση, τεχνική και οικονομική βοήθεια και στήριξη των ε, αρχών και της κυβέρνησης, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα θέσεις απασχόλησης σε τομείς που σήμερα είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης για τους νέους, τομείς με περισσότερες δυνατότητες. Και από τη μία θέλουμε να διαθέτουμε τεχνική βοήθεια, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των κυβερνήσεων για να βελτιωθεί το κλίμα το επιχειρησιακό και την ίδια ώρα να διευκολύνουμε με την διάθεση εγγύσεων να διευκολύνουμε την χρηματοδότηση για νέα σχέδια επενδύσεων κατά προτεραιότητα σχέδια και προγράμματα που υποβάλλονται από νέους στις πιο ασταθείς χώρες, στις χώρες που επικρατεί ανασφάλεια, χώρες με αδύναμη θα έλεγα διακυβέρνηση οι εγγυήσει για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για νέα προγράμματα επενδύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι το καθοριστικό. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει τους τομείς ε, προτεραιότητας, γεωργία παραδείγματος χάριν, αλλά και ο ψηφιακός τομέας. Ξέρετε ότι στην Αφρική σήμερα ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί μια νέα ελπίδα για δημιουργίες νέων θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται για νέα εργαλεία τα οποία θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα. Όσον αφορά τώρα την πολιτική μας συζήτηση, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα επεξεργαστούμε με το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών στο Business Forum μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής, θα επεξεργαστούμε το σύνορο αυτών των θεμάτων. Οι νέοι, η δημιουργία θέσεων απασχόληση, τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε και να στηρίξουμε νέες επενδύσεις. Θα δημιουργηθεί επίσης μία πλατφόρμα ανταλλαγών. Ο διάλογος αυτός λοιπόν θα ευαθυνθεί ιδιαίτερα για να προχωρήσει η κοινή πολιτική της Ευρώπης και της Αφρικής με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. Στις 30 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η συνάντηση κορυφής μεταξύ των χωρών της Αφρικανικής Υπήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν κοιτάξει κανείς την ημερήσια διάταξη και τα καθοριστικά σημεία βλέπετε ότι οι νέοι η απασχόληση των νέων, η προώθηση του επιχειρήν, η βελτίωση του διαρθρωτικού διαλόγου, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση για τους νέους. Όλα αυτά τα θέματα είναι τα θέματα προτεραιότητας αυτής της συνάντησης κορυφής. Σήμερα λοιπόν πραγματικά το θέμα μας βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής συζήτησης, βρίσκεται στην καρδιά των ανησυχιών και σαφώς θα πρέπει όλοι από κοινού να εντοπίσουμε τρόπους να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, πιο αξιοπρεπείς και πιο ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για τους νέους της Αφρικής. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ. Ερωτήσεις υπάρχουν? Η κυρία Σόιντροβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις σας. για πολλούς λόγους θα πρέπει να δράσουμε ως Ευρώπη στην Αφρική. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις, δεν θα υπάρξουν αρκετές θέσεις ε, εργασίας Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα αναμένουμε νέα μεταναστευτικά κύματα. Ένας λόγος είναι αυτό, αλλά επίσης έχουμε και μία ευθύνη ανθρώπινη και πολιτική επίσης για να δράσουμε, να επενδύσουμε, να ενισχύσουμε τις ε, κυβερνήσεις που αναφέρατε και εσείς, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τομείς όπως η εκπαίδευση κλπ. Μετά, εσείς μιλήσατε για την Αφρική ως ενωμένη ήπειρο, αλλά αυτό δεν ισχύει, δεν είναι αλήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τις διάφορες ε, χώρες που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Μπορεί εσείς ας πούμε να μας πείτε κάποια παραδείγματα εκεί όπου υπάρχουν δηλαδή πιο ευνοϊκές συνθήκες ή πιο δυσμενείς συνθήκες. Αυτό είναι ένα πρώτο μου ερώτημα. Επίσης, να πω ότι δεν αναφέρατε μια κύρια προϋπόθεση, την ειρήνη, η οποία δεν υφίσταται σε πολλές αφρικανικές χώρες ειρήνη και ελευθερία. Δεν υφίστανται σε πολλές αφρικανικές χώρες, οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα μπορούσε να δράσει πάνω σε αυτό το θέμα η Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ώστε μετά στη συνέχεια να είμαστε σε θέση να μιλάμε για εκπαίδευση κλπ. Thank Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο και για μια δεύτερη ερώτηση από την κυρία Γιουγκέριους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα της αγοράς εργασίας στην Αφρική. Ευχαριστώ που μας θυμήσατε την ε, πρώτη διακήρυξη της Φιλαδέλφειας γιατί από καιρού εις καιρών ε, έχει νόημα να ξαναγυρίζουμε στις βασικές μας αρχές οι οποίες ε, αναφέρονται άριστα στη διακήρυξη της Φιλαδέλφειας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ε, έχει να κάνει με την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών μας. Καταρχήν προς την κυρία Μοντέζη, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ είμαστε η Επιτροπή Απασχόλησης. Και πρέπει να πω ότι εκτιμώ την ε, παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιείτε. αλλά θα μπορούσατε ίσως να δείξετε, να μας πείτε σε ποιους τομείς μπορεί να βοηθήσει περισσότερο η Επιτροπή Απασχόλησης. Και το ίδιο ε, ερώτημα απευθύνω στον κύριο Κρίστιανσεν. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι ΣΔΙΤ, οι συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα που παρουσιάσατε και οι δυνατότητες που έχουν. Αλλά αν δούμε με σοβαρότητα όλα τα αριθμητικά στοιχεία, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ε, διευρύνουμε τις συμπράξεις το ταχύτερο δυνατόν γιατί η συνεργασία σας είναι καλή μεν, αλλά μπορεί να μην μπορέσουμε να φτάσουμε σε αρκετούς νέους ανθρώπους μέσα από τα προγράμματα. Τέλος, ένα τεχνικό σύστημα ε, ερώτηση προς την κυρία Σάμιουλ Όλουν Τζουβόν. μια ερώτηση που με απασχολεί πολύ. Δηλαδή, αν πάρουμε σοβαρά την σοβαρή, ε, το σοβαρό θεματολόγιο της ε, ILO για την απασχόληση και αν ε, ασχοληθούμε σοβαρά και με τις βασικές αξίες ότι δεν πρέπει μόνο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας αλλά να είναι αυτές και αξιοπρεπείς και οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας σημαίνει ότι αυτές θα συμμορφούνται προς τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ILO, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Γιατί υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το δικαίωμα του ε, οργανώνεσθε, το δικαίωμα των παιδιών που δεν πρέπει να την χάνουν εκμετάλλευσης στο, στους χώρους εργασίας. Όλα τα βασικά πρότυπα της ILO πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εδώ να τα προωθήσετε. Ίσως ε, θα έπρεπε να ε, προσθεθούν κάποια θέματα και στις γενικές διευθύνσεις και στην ILO και στα κεφάλαια που χειρίζεται. Μία ερώτηση από την κυρία Χάρκιν και μετά θα σας δώσω εσάς το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις. Στην πρώτη ομιλήτρια είπατε ότι δεν ε, έχει σημασία μόνο ο αριθμός των θέσεων εργασίας αλλά και η ποιότητά τους. Το ίδιο ισχύει και εδώ στην Ευρώπη. Για κάποιους ανθρώπους η ψηφιακή οικονομία ε, θα δώσει νέες θέσεις εργασίας κάποιες καλές. Έχουμε ομοιότητες. Μιλήσατε για το ψήφισμα του 2012 και τις τέσσερις προτεραιότητες. Μιλάμε για απασχόληση και πλούσιες θέσεις εργασίας σε περιεχόμενο. η ανάπτυξη που λαμβάνει η χώρα στην Αφρική και σε ποιο βαθμό συμβάλλει στις καλές θέσεις απασχόλησης και τι προτάσεις έχει η ILO για να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη θα δώσει καλές θέσεις απασχόλησης. Τώρα, προς τον συνάδελφο της Παγκόσμιας Τράπεζας, μιλήσατε για την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Να δούμε το τα σκέλη προσφοράς και ζήτησης παράλληλα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν ε, ε υπάρχει κάτι στο σχεδιασμό των προγραμμάτων που μπορεί να δώσει καλύτερες λύσεις αν γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Και επίσης ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει όπως αναμένετε εσείς για να υπάρξει πρόοδος προς την Κομισιόν. Αναφερθήκατε σε κάποια πολιτικά ζητήματα, αναφερθήκατε και στη μετανάστευση και για... αυτό ισχύει και για τους τρεις. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την ε, νόμιμη μετανάστευση. Ε, είναι πολύ θετικό ότι υπάρχουν συγκεκριμένα έργα ε, που προωθείται. Υπάρχει όμως δυνατότητα να επεκταθούν ή να αναβαθμιστούν γιατί παρόλο που είναι χρήσιμα και σημαντικά φαντάζομαι ότι ακόμα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν υποτιμώ την καλή δουλειά που γίνεται, από κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς, αλλά μπορεί, υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης και επέκταση. Τέλος, ακούγοντας και τους τρεις σας, ε, θεωρώ ότι έχουμε παρόμοια προβλήματα, όχι της ίδιας κλίμακας, της ίδιας έκτασης, αλλά μας απασχολούν παρόμοια προβλήματα, δηλαδή η ποιότητα της απασχόλησης, αξιοπρεπής θέσης εργασίας κλπ. Και αν δούμε την, ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω για την Αφρική, εσείς θα μου πείτε, πάντως βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι πόροι συγκεντρώνονται στα χέρια εκείνων που ήδη έχουν ε, είναι εύποροι. Αντί να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν τις θέσεις εργασίας που θέλουμε. Εσείς τι πιστεύετε, γίνεται κάτι παρόμοιο και στην Αφρική. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις μέχρι τώρα. Λοιπόν, η κυρία Σύνθια Σάμιουελ Όλον Γιουόν για να μας πει για την ILO, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια απάντηση ή κάποιο προσανατολισμό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές που έλαβαν μέρος. Εμείς επικεντρωμάστε σε τρεις τομείς, γιατί κάποια από αυτά τα θέματα διασυνδέονται. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα πολύ σημαντικό και εύγλωτο σχόλιο για την αξιοπρέπεια της εργασίας και πόσο σοβαρά το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται στην περιοχή αυτή στην Αφρική και παγκοσμίω. δύο στοιχεία να αναφέρω. Πρώτον, ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τους στόχους αεφόρου ανάπτυξης για τη μείωση ή ακόμα εξάλληψη της στόχιας αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας. Αν εμείς επικεντρωθούμε μόνο στην ποσότητα της εργασίας, τότε διατρέχουμε το κίνδυνο να έχουμε περισσότερους ανθρώπους να δουλεύουν βέβαια, αλλά να είναι φτωχοί. Να εργάζονται δηλαδή υπό συνθήκες στόχιας. Αυτό έχει επιπτώσεις και στις επενδύσεις για την κατανάλωση. Έχει επιπτώσεις στην ε, ανάπτυξη. Έχει επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση. Οπότε η οικονομικά είναι αναποτελεσματικό ή μη αποτελεσματικό να μην αντιμετωπίσει κανείς την αξιοπρεπή εργασία, τον αξιοπρεπή χαρακτήρα της εργασίας. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στο ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων αλλά η αξιοπρέπεια της εργασίας νομίζω ότι έχει μια πιο σοβαρή, μια πιο σημαντική διάσταση. Και θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι σε αυτά τα δύο ακριβώς επίπεδα θα πρέπει να ενδιαφερθούμε ως παγκόσμια κοινότητα για να διασφαλίσουμε το ότι θα προωθήσουμε πραγματικά μια αξιοπρεπή μορφή εργασίας η οποία θα συμφέρει όλους μας στο κάτω-κάτω. Επίσης, ένα άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτό που υπόθηκε σε σχέση με τις διάφορες παρεμβάσεις. Για εμάς ως Παγκοσμία Οργάνωση Εργασίας η πολυεθνική διάσταση της εργασίας θα πρέπει να αναγνωριστεί, πιστεύουμε. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Μιλάμε για την ανάπτυξη των προσόντων, των δεξιοτήτων, αλλά ανεξάρτητα με το πόσο καλές θα είναι οι πολιτικές για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα, εάν δεν υπάρχει μία αποτελεσματική συνοχή με τις εμπορικές πολιτικές, με τις πολιτικές μηχανισμού, με τις μακροοικονομικές πολιτικές, με τις πολιτικές γεωργίας, τότε δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια ολοκληρωμένη και πολυτομεακή προσέγγιση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι οι τομείς που ανέφεραν σημαντικοί, αλλά ένας τομέας κλειδί, ο οποίος είναι κρίσιμος όσον αφορά την αναβάθμιση, είναι το να διασφαλίσουμε ότι η αξιοπρεπής εργασία, ιδιαίτερα για τους νέους, νέες γυναίκες, νέους άνδρες, πρέπει να είναι ένα κύριο αναπόσπαστο στοιχείο μακροοικονομικών πολιτικών και πολιτικών εθνικής ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να καταστεί κύριο στοιχείο και τομεακών πολιτικών. Και πρέπει να σας πω ότι κάποιες παρεμβάσεις που είχαμε και πρωτοβουλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν να εστιάζουν σε αυτό. Η ιδιωτική επένδυση και οι προτάσεις που δεχόμαστε σε ποιο βαθμό εξετάζουν αυτές τις ε, παραμέτρους. Γιατί νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τομείς κλειδί που θα μας βοηθήσουν στην αναβάθμιση. Υπήρξε μια ερώτηση για το πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τις ε, προκλήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό αποτελεί και μια ευκαιρία αν την εκμεταλλευτούμε. Καταρχάς, με το να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η πρόκληση είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Δηλαδή, είναι μια πρόκληση για όλους. Όπως και οι ευκαιρίες όταν υπάρχουν είναι για όλους. Και εντάξει, τώρα εμεί εξετάζουμε την Αφρική, επειδή ακριβώ εκεί οι προκλήσει είναι πιο έντονε. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Δηλαδή, οι προκλήσει αυτέ σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου θα πρέπει να αποτελέσουν στόχευση παγκόσμια παρέμβαση, ώστε στο τέλος αυτά που λέγαμε ήδη από το 45 να γίνουν αντί μια απειλή, κάτι το θετικό. Γιατί θεωρώ ότι η φτώχεια αποτελεί ένα στοιχείο απειλής της ευημερίας παντού, όχι μόνο στην Αφρική αλλά και, αλλούς, και σε άλλες χώρες. Να το συνδέσω αυτό μάλιστα και με το στοιχείο της ε, αυξανόμενης ανισότητας. Δεν είναι μόνο θέμα που αφορά την Ευρώπη αυτό. Δεν είναι θέμα που αφορά μόνο την γεωπολιτική. Εμείς βρίσκουμε ότι στην ανισότητα η οποία αυξάνεται εντό περιφερειών και εδώ μιλάμε εντάξει για την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, αλλά και εντό χωρών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας πέρσι για την ανισότητα. Πολλές χώρες στη Νότια Αφρική είχαν σημαντικές αυξήσεις στο επίπεδο ανισότητας. Και αυτό έχει επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή βεβαίως, έχει επιπτώσεις στην ειρήνη, έχει επιπτώσεις στην σταθερότητα και βεβαίως έχει επιπτώσεις στις συνθήκες κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό είναι η συνταγή για αυτό που βλέπουμε, που παρατηρούμε ως αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση σε αυτή την Ήπειρο και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω. Εμείς εξετάζουμε την ποιότητα των θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Εμείς θεωρούμε την επιχειρηματικότητα ως ένα συστατικό. Επιχειρηματικότητα όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερους, μάλλον αν έχουμε επιχειρηματικότητα που σημαίνει ότι θα πρέπει να εντάξουμε όλο και περισσότερο στην επίσημη οικονομία, αυτό είναι μονόπλευρο. Γιατί η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας θα έπρεπε να μας βοηθάει να εντοπίσουμε τις επιχειρήσεις που έχουν παγκόσμια έφεση και να τις βοηθήσουμε, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο δηλαδή, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία που θα ήθελα να αναφέρω, αλλά θα τα αφήσω για τους υπόλοιπους ε, εισηγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Ο κύριος Κρίστιασεν τώρα. Ναι, ευχαριστώ για το πρώτο ερώτημα. Είναι διαφοροποιημένες και η Αφρική και η Ευρώπη. Μπορεί κανείς ε, να μιλήσει για τις διάφορες πτυχές αυτής της πολυμορφίας. Ποια είναι όμως τα κοινά και τα κοινά όσον αφορά την απασχόληση είναι το θέμα της παραγωγικότητας. Αυτό είναι μια πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες. Το θέμα της παραγωγικότητας πρόκειται για ένα τομέα που απασχολεί πολλούς, απασχολεί τους νέους ιδιαίτερα γιατί οτιδήποτε δεν μπορεί να παραχθεί αποτελεσματικά και με τρόπο που να συμφέρει τη χώρα εισάγεται. Υπάρχουν λοιπόν προκλήσεις στον τομέα αυτό της παραγωγικότητας διαφορετικές, αλλά είναι ένα κοινό θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες της Αφρικής. Υπάρχει βεβαίως και ο πιο παραδοσιακός τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα της απασχόλησης, στη γεωργία παραδείγματος χάρη. Υπάρχει όμως και μια κοινή δυσκολία που είναι η παροχή τροφής, ειδών διατροφής για τις αστικές περιοχές. Η Αφρική, η οποία γνωρίζει μεγάλη αστική ανάπτυξη, σαφώς και θα έχει όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για την προμήθεια ιδιών διατροφής ε, σε αυτές τις μεγάλες πόλεις και τις αστικές περιοχές. Και υπάρχουν ε, πολιτικές, ε, υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι να προμηθεθούν στην Μοζαμβίκη αλλά και αλλού είδη διατροφής, αγροτικά προϊόντα, και να καλύψουν τις ανάγκες των μεγάλων πόλεων και των αστικών περιοχών. Και βεβαίως όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν όλες τις αφρικανικές χώρες. Πρέπει να συζητηθούν, να βρεθούν λύσεις προσαρμοσμένες που να ανταποκρίνονται στα προβλήματα και στις ανάγκες. Και αυτό είναι μια πρόκληση που θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να τις αντιμετωπίσουν. Στο δεύτερο σημείο μια επιτροπή όπως αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμόδια για θέματα απασχόλησης πώς μπορεί να βοηθήσει, πώς μπορεί να συνεισφέρει. Νομίζω ότι η τελευταία ερώτηση ήταν αυτή. Μιλήσατε επίσης για κάτι το προφανές, το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Αυτό είναι ένας τρόπος συνεισφοράς. Οι νέοι στην Αφρική και όλοι αυτοί που θέλουν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσεις. Σήμερα υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν θέματα κάλυψης αναγκών της αγοράς εργασίας. Μπορεί να μην είναι ε, πολιτικά ορθό να μιλήσει κανείς γι' αυτό, αλλά η Γερμανία παραδείγματο χάρη έχει ανάγκες που δεν καλύπτονται. Και από την άλλη η μαζική στροή μεταναστών είναι κάτι που προκαλεί ανησυχίες. Η ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων όταν φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ε, γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως η 20 που φυσικά και αντιμετωπίζουν ε, τις ε, δυσκολίες αυτές, επεξεργάζονται τα θέματα της νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας, της ενσωμάτωσης των νόμιμων μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης. Και βεβαίως οι καλές πρακτικές, η ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό το μοντέλο που λειτουργεί σε μια χώρα να μπορεί να εφαρμοστεί και να μεταφορθεί και σε άλλες, είναι ιδέες τις οποίες θα πρέπει να γενικεύσουμε και να υιοθετήσουμε. Το θέμα των εμπορικών συναλλαγών, εάν δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία ε, των πολιτών μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Αν δεν μπορούν να καταργηθούν τα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, τότε η χρηματοδότηση της Ευρώπης θα πρέπει να μεταφερθεί, να στηρίξει, να πάει στην Αφρική. Και αυτό αποτελεί τμήμα της ε, πολιτικής μας για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από μικρές κινήσεις και μετά ακολουθεί μια ολόκληρη σειρά πρωτοβουλειών. Τέλος, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων και ποια είναι αυτά που έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τις α, ανησυχίες σας για το αν είναι αποτελεσματική και ολοκληρωμένη η προσέγγισή μας. Αλλά από τη μία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το μακροοικονομικό επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο, οι μεμονωμένες δράσεις και κάποιες περιοχές που πρέπει να ενσωματωθούν στα προγράμματα αυτά που λειτουργούν κάπου αλλού θα πρέπει να αναλύσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών, των τομέων, τι προσόντα χρειάζονται, τι δεξιότητες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επιτόπου δημιουργούν τις προϋποθέσεις και θα πρέπει να στηρίξουμε τις πλατφόρμες αυτές που υπάρχουν, που λειτουργούν μεταξύ των παραγωγών, μεταξύ του εργατικού δυναμικού, μεταξύ των φορέων και μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι ε, κάτι που εμείς ξέρουμε να κατευθύνουμε και συμφωνώ μαζί σας ότι τα συστήματα τα οποία λειτουργούν θα πρέπει να γενικευτούν, θα πρέπει να μεταφερθούν και αλλού. Και όσο προχωράμε μαθαίνουμε από την εμπειρία μας και βλέπουμε τι λειτουργήσε και τι απέτυχε. Ένα τελευταίο σημείο. Πιστεύω ότι μια σημαντική απειλή είναι η επέκταση της οικολογικής ευαισθησίας σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ανισότητες μεταξύ των χωρών, μεταξύ των περιοχών. Και σε κάθε περίπτωση όλοι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα υγιές οικοσύστημα και ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, ότι χρειάζεται πρόσβαση όλων στις νέες τεχνολογίες και στις νέες δυνατότητες και ότι σίγουρα θα πρέπει να μεωθεί το χάσμα και να μην αυξηθούν οι ανισότητες που ήδη υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε τον ε, λόγο στην κυρία Καλαμοντέζη από την Κομισιόν σε δύο λεπτά αναφέρθηκε και το εμπόριο που μπορεί να δώσει πολλά καλά αποτελέσματα και οι εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία δύο-τρία χρόνια προχώρησαν πολύ και με την Αφρική και με άλλα μέρη του κόσμου. Και εκεί δεν περιοριζόμαστε μόνο στις συναλλαγές με εμπορεύματα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό και όταν μιλήσουμε για, και θα μιλήσουμε και για τη γεωργία επίσης, επίσης την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφές στην Ανατολική Αφρική όπου υπάρχουν τεράστια προβλήματα τι μπορούμε να κάνουμε μαζί ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική για αυτά και βέβαια και οι νέες τεχνολογίες και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τρίτο σημείο στο θεματολόγιό μας. είναι ε, σημαντική η ψηφιακή εξέλιξη στην, ε, σε ορισμένε περιοχές της Αφρικής. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να ωφεληθούμε και εμείς και η Αφρική. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Γι' αυτό που ακούσαμε για την ε, ελευθερία και την ειρήνη και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Όπως είπε και ο Λουκ, η κατάσταση ποικίλει στο εσωτερικό των χωρών, ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης, και οικονομικής μεγέθυνσης. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου υπάρχει κατάσταση πολιτικής αστάθειας, υπάρχει έλλειψη ασφάλειας και αυτό είναι ο κύριος στόχος μας, δηλαδή να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς αυτούς. Οπότε η στήριξη της Ένωσης ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Και εγώ μόλις γύρισα από, το βορειοανατολικό κομμάτι της, ε, του Νίγηρα, όπου ξέρετε ότι έχουμε την Μπόκο Χαράμ, αυτή την οργάνωση. Ξεκίνησε από εκεί αυτή η οργάνωση τη στιγμή που αυτή η χώρα είχε τεράστιες πιθανότητες ανάπτυξης με πολλά εκατομμύρια κατοίκους και βλέπουμε ότι εκεί ακριβώς που είναι η καρδιά της γεωργικής παραγωγής, τα πάντα έχουν σταματήσει ακριβώς λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων και της εισβολής της Μπόκο Χαράμ. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα παρέμβαση μας εκεί είναι ακριβώς να στηρίξουμε τις προσπάθειες για πάυση των σειράξεων και να στηρίξουμε βεβαίω τους κύριους τομείς όπως εδώ η Γεωργία ώστε τελικά να πετύχουμε αυτή τη διασύνδεση ειρήνη-ασφάλεια και ασφάλεια-ανάπτυξη. Αλλά για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας και άλλα βασικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την οικονομική, για την ανθέρμανση της οικονομίας ή για την διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας ή την ίδια την ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν περιοριζόμαστε μόνο στις βασικές ανάγκες, Θέλουμε από τώρα να δούμε το πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ενδεχομένως την επαγγελματική κατάρτιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε προσφυγικούς ε, καταβλισμούς ώστε να ενταχθούν σε κάποιες οικονομικές δραστηριότητες. Αλλά βέβαια σήμερα οι κίνδυνοι είναι πολλαπλή στην ε, Αφρικανική Ήπειρο. Οπότε τι μπορούν να κάνουν τα κοινοβούλια ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου. Το ανέφερε και ο Λουκ Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να επιμένουμε για τον ρόλο των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Για την ανάγκη συνέχιση επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην πραγματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση κλπ. Είναι αλήθεια ότι από μόνο του ίσως αυτό να μην, έχει, να μην λέει τα πάντα, αλλά παραμένει πολύ σημαντικό και στην πολιτική ανάπτυξή μας έχουμε κάνει κάποια μετατόπιση. Έχουμε τα τελευταία χρόνια λιγάκι απομακρυνθεί από την εκπαίδευση και δώσαμε προτεραιότητα σε άλλες παρεμβάσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι συνεχίζει να παραμένει μια προτεραιότητα σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, στην Αφρική, ώστε ακριβώς να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και νομίζω ότι αυτό είπε και η διάσκεψη στο Γκέτεμπορκ το, το Σαββατοκυριακό ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και να τονίσουμε την ανάγκη της εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα αφορά τη μετανάστευση. Σήμερα υπάρχουν δυνάμεις στις κυβερνήσεις μας και στην κοινωνία των πολιτών μας που στοχεύουν στο να μετατοπίσουν την προτεραιότητα προς τη μετανάστευση, προς την αντίθεση στη μετανάστευση δηλαδή στο σύνολό τη, είτε είναι νόμιμη είτε παράνομη. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μας σφαιρικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να περάσουμε από την απασχόληση στην Ευρώπη στην απασχόληση στην Αφρικανική Ήπειρο. Και θα πρέπει δηλαδή να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα της μετανάστευσης στην Μεσόγειο μέσω μιας νόμιμης μετανάστευσης που θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πιο επικοτομητική επαφή και διάλογο με τους εταίρους μας στην Αφρικανική Ήπειρο. Νομίζω λοιπόν ο σημαντικός ρόλος του Κοινοβουλίου μπορεί να συνίσταται στο να αντιτασσόμαστε σε κάποιες σημαντικές φωνές πίεση στην Ευρώπη που είναι κατά της μετανάστευσης και σήμερα είναι κατά της μετανάστευσης στο σύνολό της, είτε είναι νόμιμη είτε παράνομη. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε διαφορετική προσέγγιση για την νόμιμη μετανάστευση και αυτό θα πρέπει να το μεταφέρουμε στο διάλογο μας με τις χώρες εταίρους μας. Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφέρθηκε. Ένα μικρό παράδειγμα έδωσα για τον Ήγηρα. για το πώς δηλαδή σήμερα προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δηλαδή, το να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, πέτυχε, μάλλον χρησιμοποιώντας το σύνολο των παρεμβάσεων και των πολιτικών μας. Δηλαδή, παρεμβάσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο εκπαίδευσης, παρεμβάσεις σε τεχνικό ακόμα επίπεδο, ας πούμε στη γεωργία και κοινωνικές πολιτικές. Δηλαδή πολλαπλές παρεμβάσεις και η πρόκληση συνεχίζει να εφίσταται γιατί δεν έχουμε μαγικές λύσεις. Έχουμε δηλαδή ένα σημαντικό διακυβευόμενο και μια προσπάθεια σημαντική ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα καταλληλότερα προγράμματα για αυτές τις παρεμβάσεις και να δούμε και ποια είναι η αξία, η αλυσίδα αξιών, ώστε να εντοπίσουμε κάποιους τομείς, ας πούμε, εντάξει, κάνουμε μια παρέμβαση στη γεωργία, αλλά στη γεωργία συγκεκριμένα σε ποιο τομέα αυτή τη αλυσίδα θα πρέπει να παρενέβω ώστε πραγματικά να κάνω μια αποτελεσματική παρέμβαση, ώστε να δημιουργήσω θέσει εργασία και οι θέσει εργασία αυτή να είναι αξιοπρεπείς για τις εμπορικές συμφωνίες τώρα, όντως αργαστήκαμε πολύ, αλλά δυστυχώς για την Αφρικανική Ήπειρο δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις οικονομικές εταιρικές σχέσεις. Στην Ανατολική Αφρική νομίζω Μαυριτανία και Νιγηρία δεν έχουν επικυρώσει ακόμα τις εμπορικές συμφωνίες και η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε με κάποιες χώρες εταίρους είναι να τους αποδείξουμε ότι έχουν πλεονεκτήματα αυτές τις συμφωνίες οικονομικά για αυτές τις χώρες για την υλοποίηση αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ακόμα χρόνο, χρειαζόμαστε ενδεχομένω και μελέτες ώστε να πείσουμε αυτές τις χώρες ότι η υπογραφή αυτών των συμφωνιών παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα για τις οικονομίες τους άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή που αποτελεί μια πολύ σημαντική πολιτική και είναι ένα στοιχείο πολιτικής για το οποίο σήμερα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το mainstreaming. Δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε παρεμβάσεις στον τομέα της Γεωργίας λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στο κλίμα από αυτές τις παρεμβάσεις στη Γεωργία. Ας πούμε, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις γεωργικές τεχνικές ώστε αυτές να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να αντιμετωπίζουμε σωστά την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή που σήμερα έχει τεράστια σημασία, ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να αναλυθεί νομίζω με τρόπο οριζόντιο πια, δηλαδή στο σύνολο των ε, δράσεών μας και μάλιστα και των δράσεών μας στον τομέα της ε, γεωργίας όπως είπαμε και σήμερα. Mm-hmm. Γεωργία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για δημιουργία θέσεων εργασίας όσον αφορά την Αφρικανική Ήπειρο. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συζήτηση, θα έλεγα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας που ξεκινήσαμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και βεβαίως οι δικές σας προτεραιότητες, η δική σας ημαρήσια διάταξη είναι πολύ συναφής με τη δική μας. Αξιοπρεπής εργασία, αυτό είναι για μας το α και το ω Μας ενδιαφέρει βεβαίως και ο κόσμος εκτός Βρυξελών. Γι' αυτό και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για την διαθεσιμότητά σας, για το ότι συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα τις επαφές μας για να μπορέσουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε από κοντά το τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές του κόσμου όπως η γειτονική μας Ήπειρος, η Αφρική. Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι δεν κάνουμε σωστά. Θα σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.